Witam Państwa. Bardzo proszę. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Ούτως ή άλλως έχουμε καθυστερήσει, ας μην το αναβάλουμε λοιπόν, ας εγκρίνουμε πρώτα την ημερήσια διάταξη. Όπως ξέρετε, έχουν γίνει πολλές αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Σας στείλαμε την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Θα μας παρουσιάσει καταρχήν η κυρία Τελαέ την ε, έκθεση γνωμοδότησή της, που ήταν αρχικά το σημείο 15 για τα αλκοολούχα ποτά, ε, σε αντικατάσταση του σημείου 5 της γνωμοδότησης ε, Σάνι για τον προπολογισμό που θα βρει το απόγευμα. Επίση, αύριο το πρωί η κυρία Πετήρ θα μα υποβάλει το σχέδιο γνωμοδότησή τη για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και όχι το απόγευμα, αλλά το πρωί. Το απόγευμα θα έχουμε τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατέτηση της Επιτροπής μας για την κατεξοδότηση πράξη για τον Ίνο ε, και η ψηφοφορία του σημείου 10 που κανονικά προβλεπόταν για το πρωί για το Ίνο για το ε, Ίνο και την αναβολή της, ψηφοφο... της κατεξοδότησης πράξης, αυτό θα μεταβεί για το απόγευμα. Ε, Οπότε είναι λογικό να ακούσουμε πρώτα το πρωί την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ινωτεράν και το απόγευμα να ψηφίσουμε για την δίμηνη αναβολή, η παράταση τη προθεσμίας κατά ένα δίμηνο. Αυτά, αυτές είναι οι αλλαγές. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσει για τις τροποποίησεις τη ημέρης διάταξη. διάταξης την δεχόμαστε. Έχουμε διερμηνία σε 16 γλώσσε. και το πρώτο σημείο είναι η εφαρμογή της ΚΑΠ και η παροχή ευελιξίας στα κράτη-μέλη, κατάσταση και προοπτικές. Και παρουσίαση θα γίνει από την κυρία Ιντατελόν, κύριε Μάλλον, από το Πανεπιστήμιο Βάγκενιγκεν και τον κύριο Τόμας Κουμόναν από το Augurix OI της Φιλανδίας. Η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Γεωργίας, ε, ζήτησε την εκπόνηση της μελέτης αυτής ε, που την ανέθεσε και τη διαχειρίζεται το Τμήμα Πολιτικής Β. Οπότε θα ξεκινήσουμε με την παρουσίαση από τους εμπειρογνώμονες, από τους εμπειρογνώμονες μας. Πρόκειται για μελέτη που είναι κοινό πόνιμα δύο φορέων, δύο ερευνητικών Ινστιτούτων. Και το θέμα είναι η παροχή ευελιξίας στα κράτη-μέλη για την εφαρμογή της κοινή γεωργικής πολιτικής. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους εμπειρογνώμονές μας, τον κύριο Ίντα Τερλόιν από το Πανεπιστήμιο, το Ερευνητικό Κέντρο του Βάγγενίγκεν και τον κύριο του Όμας Κούμονεν από το Ερευνητικό Φορέα της Φιλανδίας. Θα σας δώσω το λόγο. Έχετε 20 λεπτά για την παρουσίαση της μελέτης σας μπορείτε να κατανείμετε αυτό το 20 λεπτό όπως κρίνετε σκόπιμο μεταξύ σας. 20 λεπτά συνολικά για τους εμπειρογνώμονες για την παρουσία της μελέτης. Θα ακολουθήσει η συζήτηση με την υποβολή ερωτήσεων από τους ευρωβουλευτές. Καλωσορίζω και πάλι θερμότητα τους εμπειρογνώμονες μας και τους δίνω αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να παρουσιάσουμε τη μελέτη αυτή όσον αφορά την ευελιξία στα κράτη-μέλη στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής. Έχουμε έξι βασικά σημεία στην παρουσίασή μας. Καταρχάς θα δούμε τι εστί ευελιξία, τι αφορά. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο η ευελιξία εφαρμόζεται στα πλαίσια των άμεσων ενισχύσεων της κοινή γεωργικής πολιτικής για την περίοδο 2014-2020, θα αναφερθούμε στη συνέχεια στα εθνικά καθεστώτα ευελιξίας. Θα συζητήσουμε τη συνεχεία της επιπτώσεις της ευελιξίας για την κοινή γεωργική πολιτική, για τους στόχους της πολιτικής αυτής, για τις θεσμικές διαδικασίες και για την εφαρμογή της πολιτικής. Εν συνεχεία, ως πέμπτο σημείο, θα συζητήσουμε διάφορα σενάρια ευελιξίας, ιδίως για το μέλλον, για τις μελλοντικέ περιόδους δηλαδή της κοινή γεωργικής πολιτικής και θα καταλήξουμε έπειτα σε κάποια συμπεράσματα. Καταρχάς λοιπόν, τι είναι η ευελιξία. Η ευελιξία είναι ένας τρόπος εφαρμογής μιας πολιτικής έχουμε ευέλικτα μέτρα εφαρμογής τα οποία αφήνουν περιθώριο προσαρμογής κάποιων πολιτικών και μέτρων σε εθνικό επίπεδο. Κατά αυτόν τον τρόπο τα κράτη-μέλη μπορούν να προσαρμόσουν μια πολιτική σε συγκεκριμένε γεωγραφικές ιδιαιτερότητες ή σε συγκεκριμένε συνθήκες που μπορεί να ισχύουν στον τομέα της γεωργίας και έπειτα έχουμε και την ομοιόμορφη εφαρμογή των μέτρων όπου έχουμε ουσιαστικά κοινέ και ομοιόμορφες οδηγίες για την εφαρμογή μιας συγκεκριμένη πολιτικής. Και ποια μέτρα τώρα της κοινή γεωργικής πολιτικής χρησιμοποιείται η ευελιξία. Είδαμε ότι ε, μπορούμε να έχουμε μέτρα τα οποία αφορούν την κοινή οργάνωση αγοράς. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται ομοιόμορφα πάντα. Ξέρετε εδώ πέρα ότι έχουμε την ιδιωτική αποθήκευση, έχουμε τις ε, παρεμβατικές τιμές από τα κράτη-μέλη και διάφορες άλλες ε, τέτοιες πολιτικές. Από την άλλη έχουμε μέτρα τα οποία μπορούν να εφαρμόζονται ευέλικτα και έχουν να κάνουν κυρίως με τις ενισχύσεις και τις επιδοτήσεις προς τους γεωργούς. Αποτελούν τμήμα της πολιτικής για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τμήμα της πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου και αναφέρονται στον πρώτο πυλώνα με τις άμεσες ενισχύσεις της κοινή γεωργικής πολιτικής. Η ευελιξία έχει χρησιμοποιηθεί στην γεωργική διαθροτική πολιτική με τις πρώτες κοινωνικονομικές οδηγίες της δεκαετίας του 1970, όπου Ουσιαστικά ήδη από τότε είδαμε ότι μπορούσε ένας βαθμός ευελιξίας να χρησιμοποιείται και στο πλαίσιο της κοινή γεωργική πολιτικής. Εμείς διακρίνουμε τρεις μορφές ευελιξίας Πρώτον, έχουμε την ευελιξία ως προς την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων. Αυτό δίνει ένα περιθώριο ευελιξία, μια διακριτική ευχαίρεια στα κράτη-μέλη για την έγκριση συγκεκριμένων μέτρων. Έπειτα, έχουμε την ευελιξία ως προς τη στοχοθέτηση και ως προς το σχεδιασμό. Ουσιαστικά εδώ πέρα υπάρχει μια ευελιξία για τα κράτη-μέλη προκειμένου να καθορίσουν αυτά το επίπεδο εφαρμογής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ή τους συντελεστές ενίσχυσης για ένα συγκεκριμένο μέτρο και τέλος έχουμε τη λεγόμενη χρηματοπιστωτική ευελιξία, όπου δίνουμε ουσιαστικά το παίρνει ευελιξία στα κράτη-μέλη προκειμένου να έχουν μια περιορισμένη ανακατανομή των πόρων μεταξύ διαφόρων μέτρων και μεταξύ των πυλώνων. Ας περάσω τώρα στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασής μου που έχει να κάνει με την ευελιξία στην κοινή γεωργική πολιτική και συγκεκριμένα στις άμεσες ενισχύσεις. Θα αναφερθώ καταρχάς στη θέση των θεσμικών οργάνων του Συμβουλίου, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας το 2013. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν υπέρα κοινών ομοιόμορφων και εξορθολογισμένων μέτρων, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν υπέρ πιο προσαρμοσμένων στις τοπικές ιδιαιτερότητες και διαφοροποιημένων μέτρων, ενώ το Συμβούλιο βρισκόταν σε μια ενδιάμεση θέλετε, θέση, είχε διαφορετικές προσεγγίσεις. Πολλές φορές το Συμβούλιο ήταν υπέρ της ευελιξίας, άλλοτε πάλι ήταν υπέρ μιας ομοιόμορφης εφαρμογής των μέτρων. Οι διαφορετικές αυτές θέσεις των θεσμικών αυτών οργάνων έχουν να κάνουν με τις διαφορετικές προτεραιότητες των θεσμικών αυτών οργάνων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ μιας πιο ομοιόμορφης προσέγγισης, καθότι εστιάζεται περισσότερο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπώντας περισσότερο τους πολίτες ήταν ε, υπέρ μιας πιο προσαρμοσμένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, όπως ακριβώς αυτή διαμορφωνόταν και από διάφορες πολιτικές ομάδες, ενώ το Συμβούλιο εκπροσωπούσε πιο συγκεκριμένα τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Ας δούμε τώρα πώς οργανώνεται η ευελιξία στα πλαίσια της κοινή γεωρικής πολιτικής και ποια μορφή ευελιξίας έχουμε στις άμεσες ενισχύσεις. Βλέπετε ότι όσον αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση για τις άμεσες ενισχύσεις, όσον αφορά το greening, και όσον αφορά τον ορισμό του ενεργού γεωργού, έχουμε μόνο, στοχοθέ... έχουμε μόνο ευελιξίες προς στοχοθέτηση και το σχεδιασμό. Για την εσωτερική διακυβέρνηση τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία αποφασίζουν αν θα χρησιμοποιήσουν ε, εν μέρη σύγκληση, η μερική σύγκληση, η πλήρη σύγκληση. Όσον αφορά το πρασίνισμα, το greening, πάλι τα, τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία μπορούν να αποφασίσουν ποιε πρακτικές θα χρησιμοποιήσουν. Και όσον αφορά τον ορισμό του ενεργού γεωργού, πάλι τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν εδώ πέρα τον αρνητικό κατάλογο. Όσον αφορά τώρα την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων, όσον αφορά το καθεστώς κατόχου μικρής γεωργικής εκμετάλλευσης όσον αφορά τις γεωγραφικές εκείνες περιοχές για τις οποίες ισχύουν περιοριστικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο και όσον αφορά τι συνδεδεμένε ενισχύσει, έχουμε και τι τρει μορφέ ευελιξία. Ευελιξία προ την εφαρμογή, ευελιξία προ το στοχοθέτηση και το σχεδιασμό, ευελιξία όσον αφορά την χρηματοοικονομική πτυχή. Τα κράτη-μέλη λοιπόν αυτά τα οποία αποφασίζουν πώς ακριβώς θα χρησιμοποιήσουν τα μέτρα αυτά και πώς θα ανακατανύμουν τελικά και τους πόρους που τους αναλογούν στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής. Όσον αφορά το καθεστώς τώρα των νέων γεωργών, εδώ πέρα έχουμε την ευελιξία ως προς τη στοχοθέτηση και ως προς το σχεδιασμό και όσον αφορά την προοδευτική μείωση και τον καθορισμό ανώτατου ορίου έχουμε μόνο δύο μορφές ευελιξίας, αυτή που έχει να κάνει με την έγκριση συγκεκριμένων μέτρων και την ευελιξία που έχει να κάνει με τη στοχοθέτηση και το σχεδιασμό. Βλέπετε λοιπόν ότι οι μορφές ευελιξίας ποικίλουν με βάση τα μέτρα ή τις πληρωμές ενισχύσεις που συζητάμε κάθε φορά. Τώρα, ας περάσουμε στο τρίτο τμήμα της παρουσίασης. Ας δούμε πώς τα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει το καθεστώς ευελιξίας στο πλαίσιο των άμεσων ισχύσεων για την περίοδο 2014-2020. Θα αναφερθώ εδώ πέρα στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης, στη συνδεδεμένη στήριξη και στην ανακατανομή και την προοδευτική μείωση. Όσον αφορά τις βασικές ενισχύσεις, στην τρέχουσα περίοδο βλέπουμε ότι αποτελούν μια εξέλιξη από το καθεστώς ενιαίες ενίσχυσης, το οποίο είχαμε το 2003 μέχρι 2014. Είχαμε τέσσερα μοντέλα στο παρελθόν για την εφαρμογή της ευελιξίας αυτής. Είχαμε το ιστορικό μοντέλο, όπου οι ενισχύσεις βασικά βασίζονταν σε μια ιστορική αναφορά. Είχαμε το περιφερειακό μοντέλο, όπου είχαμε ουσιαστικά μία καταποκοπή ενίσχυση αναεκτάριο, είχαμε το μεικτό μοντέλο, όπου η πληρωμή εν μέρη βασιζόταν σε ιστορική αναφορά και εν μέρη σε καταποκοπή ενίσχυση αναεκτάριο και τέλος είχαμε το καθεστώς ενιαίας δραματικής ενίσχυσης για τα νέα κράτη-μέλη όμως μόνο. Τώρα, στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, όπου έχουμε το καθεστώς βασικής ενίσχυσης πλέον, μπορούμε να πούμε ότι το ιστορικό μοντέλο εκπροσωπείται ουσιαστικά από ένα καθεστώς μερικής σύγκλησης της βασικής ενίσχυσης. Το περιφερειακό μοντέλο εμφανίζεται με τη μορφή της πλήρους σύγκλησης από το 2015 και μετά. Το μεικτό μοντέλο αντιστοιχεί σε μια πλήρη σύγκληση αυτή προβλέπεται για το 2019, ενώ το καθεστώς ενιαίας τερματικής ενίσχυσης παραμένει το ίδιο με αυτό το οποίο είχαμε στην προηγούμενη περίοδο, 2003 με 2014 δηλαδή. Τώρα ας δούμε αν τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν το ίδιο μοντέλο κάθε φορά που μιλάμε για καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης ή για καθεστώς βασικής ενίσχυσης. Είδαμε ότι η προσέγγιση των κρατών μελών δεν ήταν πάντα η ίδια. ηταν παντα ιδια εχουμε 7 κράτη-μέλη τα οποία χρησιμοποίησαν το ιστορικό μοντέλο το οποίο δυστυχεί σε μία εν μέρη σύγκληση όσον αφορά το καθεστώς βασικής ενίσχυσης Τέσσερα κράτη-μέλη χρησιμοποιούσαν το ιστορικό μοντέλο, αλλά πέρασαν στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού σε μια πλήρη σύγκληση με χρονικό ορίζοντα το 2019. Εντοπίσαμε εννιά νέα κράτη-μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το καθεστώς ενιαίας δραματικής ενίσχυσης και στις δύο περιόδους προγραμματισμού και είχαμε και εννια κράτη-μέλη τα οποία είχαν διαφορετικό διαφορετικό σημείο αφετηρίας για την περίοδο 2003-2014 και κατέληξαν τελικά σε διαφορετικές πολιτικές στο πλαίσιο της νέας περίοδου προγραμματισμού. Η μετάβαση αυτή σε διαφορετικά μοντέλα από τη μία περίοδο στην άλλη καταδεικνύει τελικά ότι μπορούμε να έχουμε ένα κοινό σημείο κίνηση σε μια συγκεκριμένη περίοδο προγραμματισμού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε και το ίδιο σημείο άφηξη στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Μπορεί ορισμένα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν ε, με ακριβώ την ίδια προσέγγιση, αλλά να καταλήξουν σε μια διαφορετική προσέγγιση, καθώς αλλάζουμε περίοδο προγραμματισμού. Α δούμε τώρα πώς έχουν εφαρμοστεί τα μοντέλα ευελιξία όσον αφορά τη στεδεμένη υποστήριξη την περίοδο 2010-2014 βλέπετε τα κράτη-μέλη αυτά πάνω αριστερά, τα οποία χρησιμοποίησαν στεδεμένη υποστήριξη στην προηγούμενη περίοδο και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν και στην τρέχουσα περίοδο. Στη συνέχεια βλέπουμε έξι κράτη-μέλη, τα οποία χρησιμοποίησαν στο παρελθόν δεμένη υποστήριξη και στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού αποφάσισαν να μάλλον ενώ δεν χρησιμοποιούσαν, με συγχωρείτε, τη στεδεμένη υποστήριξη στην προηγούμενη, τρέχουσα περίοδο, στην προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού, στην τρέχουσα περίοδο αποφάσισαν να τη χρησιμοποιήσουν όπως το Λουξεμβούργο. Έχουμε έπειτα την αναδιανεμητική ενίσχυση. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω πληρωμές από τα κράτη-μέλη ένα εκτάριο. Πέντε κράτη-μέλη χρησιμοποιούν την εναλλακτική αυτή επιλογή. Όταν χρησιμοποιείται αυτή η αναδιανεμητική ενίσχυση, δεν είναι υποχρεωμένο το κράτος μέλος να επιβάλλει το φόρο σταδιακής μείωσης. Και αυτό ουσιαστικά έκαναν και πέντε από τα κράτη-μέλη τα οποία μελετήσαμε στην έκθεση αυτή. Όσον αφορά τώρα τα ανώτατα όρια πληρωμών ανά γεωργική εκμετάλλευση. Τα κράτη-μέλη πρέπει εδώ πέρα να χρησιμοποιούν ένα φόρο προδευτικής μείωσης για τις εκμεταλλεύσεις εκείνες οι οποίες λαμβάνουν ε, τα ανώτατα όρια πληρωμών. Τα περισσότερα κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν ένα φόρο προδευτικής μείωσης ε, της τάξης του 5% για ποσά τα οποία υπερβαίνανε τα 150.000 ευρώ αναγιορική εκμετάλλευση. Έξι κράτη-μέλη όμως χρησιμοποίησαν το ανώτατο όριο αυτό χωρίς να χρησιμοποιήσουν το φόρο προδευτικής μείωσης ενώ άλλα κράτη-μέλη, όπως βλέπετε στη διαφάνεια, χρησιμοποίησαν διαφορετικά ποσοστά προοδευτικής μείωσης με βάση το ανώτατο όριο πληρωμών το οποίο προβλεπόταν κάθε φορά. Ουσιαστικά, εδώ πέρα βλέπουμε ότι η προοδευτική μείωση δεν αποτελεί ζήτημα για τα περισσότερα κράτη-μέλη, γιατί ελάχιστε είναι οι οι οποίε επηρεάζονται από την διάταξη αυτή περί προοδευτικής μείωση. Περνώντα τώρα στο τέταρτο τμήμα τη ε, παρουσίαση αυτή, εξετάσουμε τις συνέπειες της ευελιξίας για τους στόχους πολιτικής της κοινή τουρκικής πολιτικής όσον αφορά τις θεσμικές διαδικασίες και όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα εξετάσαμε τους συγκεκριμένους στόχους της κοινή γεωργικής πολιτικής ξεκινώντας με τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων Επηρεάζεται άραγε από την ε, ευελιξία. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θέσαμε στα πλαίσια της μελέτης. Όσον αφορά τα μέτρα της κοινή οργάνωσης αγοράς, εδώ υπάρχει απουσία ευελιξίας όπως είδαμε νωρίτερα. Το ίδιο ισχύει και για το πρασίνισμα, τον οικολογικό προσανατολισμό. Κατά αυτόν τον τρόπο διατηρείται ένα ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού ανάμεσα στα κράτη-μέλη και η υποχρεωτική ενίσχυση για τους νέους γεωργούς συμβάλλει στην ανανέωση των ε, γενεών, καθώς επίσης και στη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Από την άλλη είδαμε ότι υπάρχει ένα καθεστώς ευελιξίας όσον αφορά διαφορετικές αδυναμίες μπορεί να υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο. Κατά αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στο να έχουμε βιώσιμες ε, τοπικές τροφικές αλυσίδες, αλλά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια καθυστέρηση όσον αφορά την ανάπτυξη της παραγωγικότητας. Ο δεύτερος στόχος της κοινή γεωργικής πολιτικής έχει να κάνει με τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, καθώς επίσης και με τη δράση για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Η ευελιξία που έχουμε εδώ πέρα προς τη στοχοθέτηση και το σχεδιασμό μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τα διαφορετικά πλαίσια τα οποία μπορεί να προκύπτουν από τη μία χώρα στην άλλη, αλλά μπορεί η ευελιξία αυτή να οδηγήσει σε μη αποδοτικά μέτρα. Τρίτος τώρα στόχος της κοινή γεωργικής πολιτικής, εδαφική ισορροπία. Εδώ η ευελιξία είναι σημαντική προκειμένου να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τα άνισα κατανεμημένα διαρθρωτικά και φυσικά προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουν διάφορες περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευελιξία εδώ πέρα έρχεται να υποστηρίξει τους γεωργούς και επίσης συμβάλλει στο να διατηρηθεί η δομή της αγροτικής κοινωνίας και συμβάλλει επίσης σε μια διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας. Εξετάσαμε έπειτα τις επιπτώσεις της ευελιξίας για τις θεσμικές διαδικασίες στα πλαίσια της κοινή γεωρικής πολιτικής. Επικεντρωθήκαμε εδώ πέρα στο ζήτημα της αποδοτικότητας στη διαδικασία λήψη αποφάσεων στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής και αναφερθήκαμε επίση και στο ζήτημα τη επανεθνικοποίηση τη κοινή γεωργικής πολιτική. Όσον αφορά την αποδοτικότητα τη διαδικασία λήψη αποφάσεων, είδαμε ότι η ευελιξία μα επιτρέπει να έχουμε καλύτερη προσαρμογή των μέτρων σε εθνικό επίπεδο, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε πιο διασπαρμένε, αν θέλετε, αποφάσει σε πιο, ένα πιο διασπαρμένο σύστημα λήψη αποφάσεων. Θεωρήσαμε παρόλα αυτά ότι η προσαρμογή των πολιτικών της κοινή γεωργικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο είναι μια πρακτική η οποία θα πρέπει να προωθηθεί και στο μέλλον, καθότι θεωρείται αποδοτική από το να έχουμε μια ομοιόμορφη εφαρμογή όλων των πολιτικών σε κεντρικό επίπεδο. Όσον αφορά το κίνδυνο τη επανεθνικοποίηση τη κοινή γεωργική πολιτική, όπω ξέρετε, δεν προβλέπεται κανένα βαθμό ευελιξία όσον αφορά τον πυρήνα τη κοινή γεωργική πολιτική, δηλαδή την κοινή οργάνωση γεωργικών αγορών. Από την άλλη, η ευελιξία μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές πληρωμές και ενισχύσεις με βάση την περιφέρεια ή την κατηγορία του γεωργού. Αυτό μπορεί να έχει κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στο ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού, αλλά πάντως ο κίνδυνος της επανεθνικοποίησης δεν υφίσταται Η χρησιμοποιούμενη εδώ πέρα ευελιξία αυξάνει την πολυμορφία της εφαρμογής των μέτρων της κοινή γεωργικής πολιτικής, αλλά αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί περισσότερο οριοθετημένη στοχοθέτηση και όχι επανεθνικοποίηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Όσον αφορά τώρα τις επιπτώσεις της ευελιξίας για την εφαρμογή της κοινή γεωργικής πολιτικής, τη συγκεκριμένη εφαρμογή των μέτρων, Επικεντρωθήκαμε εδώ πέρα στην πολυπλοκότητα της εφαρμογής όσον αφορά το ισότιμο επίπεδο ανταγωνισμού για όλα τα κράτη-μέλη. Είδαμε ότι η ευελιξία τελικά έρχεται να μεταθέσει την πολυπλοκότητα αυτή των μέτρων της κοινή γεωρικής πολιτικής από το κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο στο εθνικό επίπεδο. Από την άλλη, η ευελιξία σε καμία περίπτωση δεν αυξάνει η ίδια την πολυπλοκότητα των μέτρων. αν βέβαια διατηρηθεί το φυστάμενο επίπεδο στοχοθέτηση. Τώρα, όσον αφορά το ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, την ισονομία που θα πρέπει να εφίσταται ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ακριβώ επειδή δεν έχουμε ευελιξία στα μέτρα τη κοινή οργάνωση γεωργικών αγορών, το ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού τελικά δεν επηρεάζεται. Η ευελιξία όμω μπορεί να έχει κάποιε αρνητικέ συνέπειε σε συγκρίσιμες περιφέρειες, συγκρίσιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις που λαμβάνουν ε, πάνω κάτω τις ίδιες ενισχύσεις. Παρ' όλα αυτά δεν προκύπτουν κάποια απατηλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ακριβώς επειδή χρησιμοποιούμε κάποιο βαθμό ευελιξίας. Μα ζητήθηκε συνεχεία να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε κάποια σενάρια για το μέλλον της κοινής γεωκρίσης πολιτικής. Επί του παρόντος δεν προβλέπεται κανένα βαθμό ευελιξίας όσον αφορά τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την κοινή οργάνωση γεωργικών αγορών. Υπάρχει ευελιξία όσον αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου και όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις. Αυτό είναι το σενάριο παριθμών 2 που βλέπετε στη διαφάνεια και θα μπορούσαμε έπειτα να φανταστούμε και ένα σενάριο στα πλαίσια του οποίου θα είχαμε ευελιξία και για τις τρεις κατηγορίες μέτρων της κοινή γεωργικής πολιτικής αυτό είναι το σενάριο παριθμών 3. Και έπειτα έχουμε και το σενάριο εκείνο στο οποίο δεν προβλέπεται καμία απολύτως ευελιξίας, όπου έχουμε δηλαδή ομοιόμορφη εφαρμογή όλων των τριών κατηγοριών μέτρων της κοινή ζωρικής πολιτικής. Είδαμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διαφορές όσον αφορά την εφαρμογή των πολιτικών στόχων της κοινή γεωργικής πολιτικής με βάση την κατηγορία μέτρων στην οποία αναφερόμαστε, θέλαμε να δούμε αν χρησιμοποιώντα ένα συγκεκριμένο σενάριο ευελιξίας θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα τα οποία αντοπίσαμε στη μελέτη. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε φορά εμφανίζονται νέε εντάσει ή νέε τριβέ. Ας περάσουμε τώρα στις καταληκτικές μας παρατηρήσεις όσον αφορά πάντα την παροχή ευελιξίας στα κράτη-μέλη στην εφαρμογή της κοινή γεωρικής πολιτικής. Μπορούμε να πούμε ότι τα μέτρα κοινή οργάνωσης γεωργικών αγορών εφαρμόζονται ομοιόμορφα, ενώ οι άμεσες ενισχύσεις και τα μέτρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου εφαρμόζονται με ένα βαθμό ευελιξίας. Δεύτερον, το εφιστάμενο καθεστώς ευελιξίας επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα προβλήματα και το, τους επιτρέπει επίσης να πετυχαίνουν γεωγραφικά οριοθετημένους στόχους. Τρίτον, η ευελιξία αυτή δεν θα πρέπει να θεωρείται σε καμία περίπτωση ως επανεθνικοποίηση της κοινής πολιτικής, αλλά αποτελεί περισσότερο οριοθετημένη στοχοθέτηση, οι υφιστάμενες μέθοδοι ευελιξίας έχουν ε, εν γέννη περισσότερο θετικές παρά αρνητικές επιπτώσεις και τέλος καταλήγουμε στο συμπέρασμα δεν υπάρχει λόγος να τροποποιήσουμε το υφιστάμενο καθεστώς ευελιξίας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε ε, Δόκτωρ Τέρλουιν. Θα περάσουμε τώρα στη συζήτηση με Ερωτήσει και παρατηρήσει από τους ευρωβουλευτέ. Ο πρώτος που ζήτησε το λόγο είναι ο κύριος Άλμπερτ Ντες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εμπειρογνώμονές μας για την παρουσίαση της μελέτης τους. Είναι σημαντικό να γίνει διαφοροποίηση, διάκριση μεταξύ των διαφόρων πτυχών αυτού του θέματος. φάνηκε και στην τελευταία μεταρρύθμιση κάπου ότι αμελήσαμε κάποιες πτυχές και ευελιξία σημαίνει ίσως μείωση της εμβέλειας της κάπου στην Ευρώπη. Σίγουρα χρειαζόμαστε αυτήν την ευελιξία σε κάποιους τομείς, δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πολιτική για του νέου γεωργού. Σε μερικέ χώρε δεν είναι αρκετό ο αριθμό ε, των νέων γεωργών, οπότε θα πρέπει να αυξηθούν. Σε άλλε χώρε είναι μεγάλο ο αριθμό των νέων γεωργών. Τώρα έχουμε ένα κανόνα που μιλάει για μέχρι το 50%, αλλά ε, εναπόκειται στα κράτη-μέλη και μερικά είναι περισσότερο υπέρ τη ευελιξία. Και αν δούμε τη σύγκριση μεταξύ άμεσων ενισχύσεων και συνδεδεμένων ενισχύσεων, ερωτώ μήπω έτσι ε, αν έχουμε ανομοιόμορφες προσεγγίσεις και υπερβολική ευελιξία, μήπως τρευλώσουμε τελικά τον ανταγωνισμό, γιατί μερικές χώρες έχουν υψηλά επίπεδα ε, συνδεδεμένων ενισχύσεων για το βόλιο κρέας, για παράδειγμα, κάτι που δεν ισχύει σε όλες τις χώρες και άρα θα έρθουν ε, σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα η παραγωγή τους. Δεν είναι αυτό τρεύλος ανταγωνισμού. Επίσης υπάρχουν ακόμη σοβαρές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και το έχουμε ξαναπεί. Για τις άμεσες ενισχύσεις, ο παρακαθήμενος, ο κύριος Δόρφαν, ε, από το Νότιο Τυρόλο, ε, ε, λαμβάνει 17 ευρώ ένα εκτάριο ενίσχυση, ενώ σε άλλα μέρη της Ευρώπης οι γεωργοί λαμβάνουν 1000 ευρώ ένα εκτάριο. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές, δεν πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Επίσης, ακόμη και οι ιστορικές μερικές περιοχές δεν έχουν πάνω από το 50% του μέσου όρου. Θα πρέπει να φροντίσουμε να αποκατασταθεί μεγαλύτερη δικαιοσύνη και ισότητα στην Ευρώπη. Μια και τον αναφέρετε, ο κύριος Ντόρφμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συνεχίσω εκεί που σταμάτησε ο συνάδελφος Ντες. Μας είπατε ότι η ευελιξία θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Δεν είναι απλοϊκή, υπεραπλουστευμένη αυτή η διαπίστωση. Έχετε κάνει έρευνε, έχετε όντω διαπιστώσει στρέβλωση ανταγωνισμού λόγω υπερβολική ευελιξία ή όχι. Ίσως δεν είχατε την ευκαιρία λόγω του περιορισμένου χρόνου να αναπτύξετε όλες τις λεπτομέρειες μελέτη σας ή δεν προλάβατε να διαπιστώσετε τέτοια στρέβλωση. Ε, Όντω στις συνδεδεμένε ενισχύσει για το βόλιο κρέα υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των κρατών μελών και σε ό,τι αφορά το βασικό πριν. Ερωτώ λοιπόν, όντω διαπιστώσατε στρέβλωση ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών ή μπορείτε να αποκλείσετε κάτι τέτοιο. Ο κύριος Λουαζό. Ευχαριστώ. Αν κατάλαβα καλά, μιλούμε για παροχή ευελιξία στα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει και κάποιο βαθμό αυτονομία για τα κράτη-μέλη. Και φαντάζομαι θα το έχετε μετανιώσει, γιατί συνεχώ προσπαθείτε να επιβάλλετε την πολιτική σα στα κράτη-μέλη. Εγώ θεωρώ ότι η γνήσια ευελιξία ισοδυναμεί με το να αφήσουμε τα κράτη-μέλη ελεύθερα να ασκήσουν την γεωργική του πολιτική ανάλογα με τι ανάγκε τη και όχι να επιβάλλετε μέσω των οδηγιών σα τον έλεγχό σα. Για παράδειγμα, η Συμφωνία ΣΕΤΑ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης. Είπαμε, είδαμε ότι θα ε, εφαρμοστεί προσωρινά από τον επόμενο Σεπτέμβριο η συνθήκη ΣΕΤΑ με τον Καναδά. Χωρίς να έχουν λόγο οι εθνικές βουλές και χωρίς να χρειαστεί να κυρώσουν ή όχι τη συμφωνία ΣΕΤΑ. Φαίνεται ότι παρακάμπτεται ε, τα Εθνικά Κοινοβούλια και δεν είστε βέβαιοι για το αποτέλεσμα. Καλή βέβαια η δημοκρατία φαίνεται, αλλά μόνο όταν συμφωνεί κανείς μαζί σας. Αυτή είναι η δημοκρατία που έχετε στο μυαλό σας. Αυτό και αν είναι ε, λαμπρό παράδειγμα ευελιξίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντριέ. Πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και Τερίνεν για την ποιότητα της παρουσίασης και την εργασία της βλέπουμε ότι αυτή η ευελιξία χρειάζεται όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις. Και αφορά βεβαίως την ανάπτυξη της πέθρου, όπως είπατε κι εσείς. Αν λοιπόν φαίνεται λογικό να έχουμε κοινού κανόνες, αυτό θα πρέπει να αφορά και τον προπολογισμό για τη μεταρρύθμιση, ώστε να αποφύγουμε δηλαδή και τη αστρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ παραγωγών. Αυτό είναι και το δικαίωμα του προγράμματος που εφαρμόσαμε. Στη μελέτη πάντως είπατε ότι για αυτές τις πληρωμές ένα κομμάτι χρησιμοποιείται από όλες τις χώρες. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ή να προβλέψουμε περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τις ε, περιφέρειες ιδιαίτερα τις ορεινές περιφέρειες ή περιοχές όπου έχουμε συγκεκριμένες σχεδιάσεις με δραστηριότητε ε, κοινοτροφικές και τα ώστε να τους ωφελήσουν. Μετά για τον πρώτο πλέον να πω κάτι. Για τις πληρωμές, ξέρετε, έχουμε τις προποθέσει. οι τιμές, οι, οι επιφάνειες, οι κοκκέ προποθέσει και συνθήκες κτλ. ώστε να έχουμε τέλο πάντων καλύτερο έλεγχο από την Κομισιόν, αλλά δεν λαμβάνουμε υπόψη μας την ευκόλυνση των ε, γεωργών όσον αφορά το, το πρασίνισμα. Μήπως λοιπόν για το πρασίνισμα, πέρα από την βιολογική γεωργία, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και άλλα συστήματα παραγωγής βιώσιμα και αηφόρα για να διευκολύνουμε τους αγρότες. Μήπως λοιπόν χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία. Γιατί εδώ στον αφορά το πρασίνισμα ξαναλέω. Ας πούμε τι γίνεται με την πολιετή συμβατική γεωργία μέσα της οποίας ας πούμε, η γεωργία θα πρέπει να πετύχει συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά τη βιωσιμότητα και η οποία θα πρέπει να επαναξιολογείται μετά από κάποια χρόνια. Σας ευχαριστώ κύριε Σλάιερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάτι λείπει νομίζω εδώ από την ε, εισηγήση που ακούσαμε. Νομίζω ότι εντάξει αναφέρθηκα κάποια πράγματα αλλά λείπουν κάποια κέρια ζητήματα και θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται με την εφαρμογή της ευελιξίας ε, σε κάποιες χώρες, ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Στο δεύτερο πυλώνα, ας πούμε, θα μπορούσαμε και να χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλα στοιχεία επειδή έχουμε εμείς διαφορετικούς ορισμούς. Μήπως θα πρέπει να δούμε ακριβώς πώς χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία η κάθε χώρα και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ομοιόμορφη αντίληψη από τους γεωργούς στις διάφορες χώρες, ενώ αυτό δεν ισχύει. Μιας και μιλάμε για την Ευρώπη και για την γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου, είναι ξεκάθαρο θα πρέπει να εμπλακούν περισσότερο οι Γεωργία. να συμμετάσχουν περισσότερο Γεωργία μα μιλάμε για ευελιξία. Τι γίνεται λοιπόν με τα αποτελέσματα, τα αρνητικά και τα θετικά αποτελέσματα. Μήπως θα μπορούσατε να επικεντρωθείτε περισσότερο στα αποτελέσματα της ε, εφαρμογής. Είπατε ότι μπορεί να προκύψουν, να ανακύψουν τέλο πάντων εντάσεις, αλλά μπορείτε να το αναλύσετε περισσότερο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την εισηγήση. Θα ήθελα να πω το εξής. Αν δείτε πώς έχει αλλάξει η ΚΑΠ, νομίζω ότι θα μπορούσαμε πολλά να πούμε όσον αφορά την προσαρμογή των πληρωμών. Στην αρχή της διαδικασία είχαμε διαφορές εκατοντάδων ευρώ ένα εκτάριο. Προσπαθήσαμε να τα αυτεγραμμίσουμε όλα αυτά και ακολουθήσαμε ένα μοντέλο ιστορικό όπου όμως τελικά αποδεικνύεται δύσκολο να υπάρχει ισοτιμία στο μοντέλο αυτό γιατί ακριβώς υποχωρεί η ιστορικότητα αυτού του μοντέλου. Θα πρέπει λοιπόν να το αναθεωρήσουμε, να το ξαναδούμε αυτό και η ευελιξία πραγματικά είναι η λέξη κλειδί. Πρέπει να υπάρχει όμως ισοτιμία ξαναλέω, γιατί η ευελιξία νομίζω ότι δεν βοηθάει τους πάντες. Η ελαστικοποίηση λοιπόν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις καταστάσεις που ισχύουν σε διάφορες χώρες και αυτό είναι μια ασθενοπός. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε περισσότερο για το δεύτερο πυλώνα. Κάτι που ισχύει και για το οποίο λυπάμαι είναι ότι οι πληρωμέ στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα δεν βοηθούν ακριβώ στην Γεωργία, γιατί νομίζω υπερβολικέ αμοδιότητε υπάρχουν στι χώρε μέλη για τον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται αυτέ οι πληρωμέ. Θα πρέπει λοιπόν οι χώρε να είναι σε θέση να μεταφέρουν ε, πληρωμέ από το δεύτερο στον πρώτο πυλώνα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να δημιουργήσουμε ε, δυνατότητε για γεωργού. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε στην Ένωση ότι ο δεύτερο πυλώνα θα πρέπει να χρησιμοποιείται με ένα πιο στοχευμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μα απασχολήσει για το μέλλον. Ε, Επίση, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονό ότι εντάξει, οι πληρωμέ είναι ένα ζήτημα, αλλά η κάθε χώρα έχει δικούς τους κανόνες φορολογικούς, ε, κανόνες που αφορούν την ασφάλεια, την υγιεινή. Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι στόχος μας εδώ στις διάφορες χώρες θα πρέπει να είναι να υπάρχει μια εναρμόνιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακριβώς αποδεικνύει αυτή η έκθεση πόσο δύσκολο είναι να είναι ευχαριστημένοι όλοι και το τωρινό σενάριο είναι η λιγότερο κακή τέλο πάντων επιλογή με ένα κοινό παρανομαστή. Θα πρέπει λοιπόν η Ένωση να αναλάβει κάποια ευθύνη όσον αφορά τι επικρίσει τη τωρινή ΚΑΠ που είναι ιδιαίτερα περίπλοκη για του γεωργού, ιδιαίτερα στα πλαίσια προσυνείσματο, τον όρο που ακούσαμε δηλαδή, όρο ο οποίο τέλο πάντων περιπλέκεται όλο και περισσότερο και δυσκολεύει τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη μα ε, τι ε, επιπτώσει που υπάρχουν για τους γεωργούς, για τις διαφορές μεταξύ ε, νομοθεσιών και άλλων στοιχείων που αφορούν με διαφθορά κλπ. Και μάλιστα έχω κατά νου και τους δικούς μου τη στιγμή που είναι δύσκολο οι δικοί μου να συμπληρώσω τέλο πάντων αυτές τις, ε, αυτά τα έγγραφα για τις ε, πυρομές. Είναι περίπλοκα. Νομίζω ότι αυτή η ισοτιμία είναι κάτι το φανταστικό, κάτι το ανύπαρκτο και νομίζω ότι στην έκθεση ακριβώς τονίζεται η ένταση, η σύγκρουση όσον αφορά την νομοθεσία και την προστασία της ατομικότητας. Θα πρέπει λοιπόν να ρωτήσω, αυτό ωφελεί αυτούς που δουλεύουν σε αυτόν τον κλάδο ή μήπω αποδεικνύει ακριβώς το πόσο κακό είναι το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να πούμε ότι θα έπρεπε να αναφέρουμε τον όρο αμοιβαία αναγνώριση. Επιτέλους, γιατί αν θέλουμε να έχουμε μετά τον Brexit ένα είδος ελευθέρου εμπορίου, ώστε η Ένωση των 27 να, έχει, να στέλνει τα φρούτα και τα κρασιά εύκολα στο Ενωμένο Βασίλειο και αντίστροφα, τότε η αμοιβαία αναγνώριση θα μπορούσε να κάνει το πολύ χρήσιμο εδώ. Να το λάβετε λοιπόν υπόψη σας. Ευχαριστώ ό,τι αφορά την πρόσληψη συμβούλων. Ε, έτσι, προσλαμβάνοντα συμβούλου, δημιουργούμε και νέε θέσει απασχόληση, αν ο κάθε χρειάζεται και το συμβουλό του. Η κυρία Μίλλερ, σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ θερμά για την παρουσίαση τη μελέτη σα. Θα ήθελα να ζητήσω μία διευκρίνηση για τις διαρθρωτικές αλλαγές. Αναφερθήκατε και σε αυτό το θέμα. Μιλήσατε για το πώς εφαρμόζεται η κοινή αγροτική πολιτική στα κράτη-μέλη και είπατε στην ουσία δεν έχουμε κοινή γεωργική πολιτική ουσιαστικά γιατί υπάρχουν τόσο διαφορετικές δυνατότητες μετά εφαρμογής της ε, ΚΑΠ που τελικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ενιαία ΚΑΠ. Μπορείτε να μας το αποδείξετε όμως αυτό με συγκεκριμένα, με αριθμητικά στοιχεία για το πόσο διαφορετικά εφαρμόζονται τα μέτρα από τα κράτη-μέλη. Γιατί κάνατε μία σύγκριση, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε πιο διεξοδικά τις διαφορές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Καταρχήν για το χαρακτηρισμό του Γιώργου, για τον ορισμό του Γιώργου Έχετε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τις ε, οικογένειες των Γεωργών. Και επίσης θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους μικροκαλλιεργητές μου λείπουν πολλά στοιχεία και έχω πολλέ απορίε για το θέμα αυτό. Κύριο Φλάναγκαν, σα ευχαριστώ. Ποια είναι η γνώμη σα ε, καταρχήν ω προ το πρόβλημα αξιοπιστία, που είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα τη κοινή γεωρικής πολιτική. Η ευελιξία θα μπορούσε να είναι θετικό στοιχείο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ε, έχουμε την περίπτωση όπου δώσε θάρρος στο χωριάτι, θα σα ανέβει στο κρεβάτι όπως λέμε. Και στην Ιρλανδία είχαμε μερικές φορές ε, ε, ευελιξία, αλλά τους δίνουμε το δάχτυλο και μας τρώνε το χέρι μερικές φορές ε, και ίσως είχαμε ανεπιθύμητα αποτελέσματα, γιατί συχνά μιλάμε για πληρωμές στα πλαίσια ενισχύσεων για δάση σε ανθρώπους που δεν είδαν ούτε τι μορφή είχε ένα αγρόκτημα και δεν είναι πραγματικά γεωργοί και παρόλα αυτά λαμβάνουν ενισχύσεις. Οπότε θα πρέπει να δούμε ε, τι συμβαίνει σε μερικές περιπτώσεις όταν παρέχουμε ευελιξία και πώς η χορήγηση αυτής της ευελιξίας υπονομεύει την ίδια την αξιοπιστία της κοινή γεωργικής πολιτικής. Επίσης, ε, μερικές φορές ε, λέμε ότι θα πρέπει να γίνουν περικοπές στην ΚΑΠ γιατί δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια λόγω και του Brexit μεταξύ άλλων. Και σε τελική ανάλυση είναι δύσκολο να, να δικαιολογήσουμε ότι δίνουμε μισό εκατομμύριο ευρώ σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία. Πέρασαν και δεν ακούπησαν. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα ως, αυτό, ε, ως προς αυτό. Επίσης αναφερθήκατε στην πολιτική ανταγωνισμού και το κατά πόσο ε, μια τέτοια ευελιξία επηρεάζει το θεμητό ανταγωνισμό. Τις προάλλες ε, είχαμε σε κοινή συζήτηση τους επιτρόπους Χόγκαν και Φερστάγκερ και είπαμε στην Επίτροπο Φερστάγκερ πώς είναι δυνατόν να εξηγήσουμε ότι ένας γεωργός λαμβάνει χίλια ευρώ ένα εκτάρι και ο γείτονάς του τίποτα απολύτως. Ε, δεν μπόρεσα να μας απαντήσει. Ε, ελπίζω ε, να ενημερωθεί η κυρία Βεστέγκερ, γιατί αν πραγματικά έχει κάποιο νόημα ανταγωνισμό, πώ είναι δυνατόν να ανταγωνιστεί κάποιον που λαμβάνει χιλιάδε ευρώ, ενώ εσύ ο ίδιο δεν παίρνει ε, ούτε ένα λεπτό. Οπότε δεν υπάρχει σίγουρα θεμητό ανταγωνισμό σε τέτοιε άνισε περιπτώσει. Ο κύριο Μπούντα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ του εμπειρογνώμονε για την παρουσίασή του. Νομίζω ότι πολλά θα διδαχθούν και οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη μελέτη αυτή, γιατί μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι οι υπάλληλοι της DG Agri είναι τελείως άσχετοι με την πραγματικότητα της γεωργίας. Είπαμε ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους γεωργούς και σίγουρα αυτή η στήριξη, αυτές οι ενισχύσεις στόχο έχουν την αύξηση της παραγωγής. Το έχω δηλώσει επανειλημμένος ότι δεν είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο μάλλον να παράγει κανείς προϊόντα. Το πιο δύσκολο πολλές φορές είναι να τα διαθέσει σε εμπορία ή να τα πουλήσει. Και δυστυχώς διαπιστώνω ότι εδώ σε πολλές προτάσεις που κάνουμε δεν σκεφτόμαστε ε, τις συνέπειες που μπορεί να έχουν. Θα πρέπει να διευκολύνουμε τους γεωργούς να διαθέτουν τα προϊόντα τους, ε, ώστε να μην είναι έρμεα των σούπερ μάρκετ, των μεγάλων αλυσίδων διανομής. Το περασμένο Σαββατοκύριακο συνάντησα αγρότες από ορεινές περιοχές της Ρουμανίας και ένας νέος γεωργός μου είπε ότι όταν ήταν 18 χρονών στο μεταξύ μεγάλος έγινε 24, αγόρασε μια αγροτική εκμετάλλευση και είπε ότι τώρα θέλει να έχει πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και παρόλο που είναι ο ίδιος νέος Γεωργός, μόλις 24 ετών, μου είπε ότι δεν έχει καμία πρόσβαση στα γεωργικά κονδύλια. Αν μιλάμε λοιπόν για ευελιξία, θα πρέπει πραγματικά να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να ορίσουν τις περιοχές που χρήζουν περαιτέρω στήριξη στη γεωργία τους. Γιατί αν έρθει κανεί από τι Βρυξέλλε και πει απλώ στα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει οι γεωργοί να λαμβάνουν ενίσχυση μέχρι τα 40 του, τότε δεν του βοηθάμε. Απλώ περιορίζουμε τα κράτη-μέλη στο περιθώριο ελιγμών του και στο πεδίο κινήσεών του. Και αυτό είναι ε, περιττό, νομίζω, και άδικο. Η κυρία Σένορα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και να υποβάλω μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αν έχει σκοπό να κάνει κάτι. Γιατί πραγματικά οι μικρές εκμεταλλεύσεις ε, είναι οι φτωχοί συγγενείς της ΚΑΠ ε, που έχουν ε, παραμεληθεί τελείως. Υπάρχει κάποια δυνατότητα να λάβουν ενισχύσεις και οι μικρές εκμεταλλεύσεις. Θα κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να μην ξεχνούν τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Γιατί αυτά τα μικρά αγροκτήματα ε, διαφυλάσσουν τις θέσεις εργασίας και επίσης ε, ε, κρατούν το πληθυσμό στην Ήπεθρο και εξασφαλίζουν την οικονομική του επιβίωση. Κάτι που είναι σημαντικό σε ζώνες όπως η Γαλλικία. Παρόλο που δεν εφαρμόζεται όντω αυτή η στήριξη στις μικρές εκμεταλλεύσεις. Ή δεν εφαρμόζεται καθόλου ή εφαρμόζεται πολύ λοιπώς. Κάτι άλλο που επίσης είναι πολύ σημαντικό είναι το ότι δεν καταφέραμε ούτε με την ευελιξία να πατάξουμε τις ανισότητες ή τις διακρίσεις στην κατανομή των ε, γεωργικών κονδύλιων μεταξύ των διαφόρων κλάδων ή μεταξύ των διαφόρων γεωργών και των διαφόρων ειδών εκμεταλλεύσεων. Πρόκειται ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλλετε προτάσεις για να αποκαταστήσετε αυτή τη δίκαιη μεταχείριση. Ευχαριστώ κύριο Δεκάστρο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους εισηγητές και του ευχαριστώ για τα συμπεράσματα. Γιατί φαίνεται ότι το όριο μεταξύ ευελιξία και παρεθνικοποίηση είναι πολύ συχνό. Οπότε, όπω είπατε και εσεί είναι καλό να μην πάμε παραπέρα. από αυτό δηλαδή που κάνουμε εδώ στην ΚΑΠ. Παρ' όλα αυτά, σε σχέση με αυτές τις ενισχύσεις, τις συνδεδεμένες, για κάποιες χώρες θα υπάρξει περισσότερη ευελιξία. Εξάλλου το οργανισμό αυτό το νόμιμο τον έχει υποβάλει η Επιτροπή μας. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό με τρόπο μη κυκλικό. Οπότε οι συνδεδεμένες πληρωμές ε, αλλάζουν φύση και δεν αφορούν τέλο πάντων την κατεύθυνση της επαρεθνικοποίησης. Μάλλον αποτελεί ένα εργαλείο παραπάνω για τις χώρε μέλη για να στηρίξουν τα εισοδήματα των γεωργών σε συγκεκριμένες χρονιές. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο, στο όμοιο, στον κανονισμό, προτείνουμε ετήσια ευελιξία. Τι άποψη έχετε γι' αυτό. Η κυρία Ράς Γκαρσία, παρακαλώ. Δεν περίμενα να μου δώσετε το λόγο τόσο γρήγορα. Ευχαριστώ πάντω. Θα ήθελα να πω ότι σε ό,τι αφορά την μελέτη και τα περιθώρια λιγμόνως προς την ευελιξία. Συμφωνώ με, κυρία, τον κύριο Δεκάστρο ότι είναι θετικά τα αποτελέσματα και ε, ως προς την αγροτική ανάπτυξη είναι αρκετά ε, ελκυστική ευελιξία για να μας επιτρέψει την υλοποίηση των στόχων της ΚΑΠ. Αλλά θα περιορίζω σε αυτό το σημείο, γιατί αν την επεκτείνουμε την ευελιξία και στα μέτρα αγοράς θα οδηγηθούμε σε πανεθνικοποίηση τη κοινή γεωργική πολιτική. Και αυτό είναι η κόκκινη γραμμή και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να την υπερβούμε. Εγώ συμφωνώ ότι τα τωρινά περιθώρια επιδέχονται κάποιε μικρέ ε, αλλαγέ και βελτιώσει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επεκτείνουμε την ευελιξία και σε άλλα μέτρα. Γιατί, επαναλαμβάνω, η επανεθνικοποίηση τη κοινή γεωργική πολιτική είναι μια κόκκινη γραμμή που σε καμία περίπτωση δεν είμαστε διατεθειμένοι να την καταπατήσουμε. Ευχαριστώ, κυρία Γιλέρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τερλάιν κάτι που δεν κατάλαβα καλά από την παρουσίαση. Κάποια στιγμή είπατε ότι είναι θετικές οι συνέπειες της ευελιξίας, γιατί μπορούν να αυξηθούν οι δαπάνες σε συγκεκριμένα θέματα. Όμως, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των στόχων της ΚΑΠ, η αξιολόγηση σας είναι θετική ως προς την ευελιξία αρνητική, γιατί με την τελευταία μεταρρύθμιση επιτρέψαμε στα κράτη-μέλη να διατηρήσουν το γεωργικό τους ε, προϋπολογισμό εξαιτίας της ε, ελαστικοποίησης των άμεσων ενισχύσεων και του δεύτερου πυλώνα, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι με την ευελιξία αυτή υλοποιούμε τους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής. Και σε, αν δεν υλοποιούμε του στόχου, θα πρέπει κάπω να τροποποιήσουμε αυτή την ευελιξία που γενικώ την κρίνατε θετικά. Όχι στη διαφεροποίηση μεταξύ των περιφερειών, γιατί σε μερικέ περιπτώσει η ευελιξία επέτρεψε σε χώρε με ιστορικά δικαιώματα να κρατήσουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο γεωργικού προπολογισμού. Δεν κατάλαβα όμω, ε, υλοποιούνται οι στόχοι τη ΚΑΠ με την ευελιξία αυτή. Γιατί εμεί έχουμε πολλά σοβαρά προβλήματα και ένα από αυτά είναι η νέοι γεωργία. Σε λίγο, ο εκπρόσωπος του Ελεκτικού Συνεδρίου θα μας παρουσιάσει την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πολιτική για τη στήριξη των νέων γεωργών είναι αναποτελεσματική και άκαρπη. Θα ήθελα λοιπόν να σταθείτε λίγο περισσότερο στους νέους και, για το, και στο κατά πόσο η, ευελιξία και η παροχή ευελιξία στα κράτη-μέλη έχει αποφέρει καρπούς ιδιαίτερα για τους νέους γεωργούς και δεν ξέρω για τους ηλικιωμένους, θέλετε να τους ε, ε, ξελείψετε, αλλά νομίζω προς τους ε, νέους γεωργούς δεν είναι εντυπωσιακά το αποτελέσμα της ευελιξίας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι όταν ακούμε όλες αυτές τις διαφορετικές παρουσιάσεις βλέπουμε τελικά και τις διαφορές που υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω ότι ε, οι περισσότεροι συναδελφοί μου θα μείνουν εκεί για την παρουσίαση του ελεκτικού συνεδρίου. Νομίζω ότι το ελεκτικό συνέδριο θα καταλήξει σε άλλα συμπεράσματα από εσά σε σχέση με την ευελιξία. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω αυτή τη στιγμή να προδικάσω τα συμπεράσματα τη έκθεση που θα ακούσουμε στο μέλλον σε λιγάκι. Το πρόβλημα είναι ότι ε, όσο περισσότερη ευελιξία έχουμε τελικά στα κράτη-μέλη, τόσο πιο δύσκολο θα είναι για το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, αλλά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να επαληθεύσει τελικά αν όντως τα ευρωπαϊκά κονδύλια χρησιμοποιούνται με τρόπο αποτελεσματικό και στοχοθετημένο και αν τελικά όντως οι βασικοί στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής επιτυγχάνονται. Και αυτό διότι, όπως ξέρετε και το ακούσαμε, δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι ορισμοί σε επίπεδο κρατών μελών. Και επειδή πολύ συχνά επικεντρώνουμε τελικά πάρα πολλούς σπόρους στο να δούμε τελικά αν έχουμε επιτύχει ή όχι τους στόχους μας, ενώ ένα μεγάλο τμήμα του κοινοτικού προπολογισμού δαπανάται, χωρίς τελικά να έχουμε στο τέλος συγκεκριμένες πληροφορίες στα χέρια μας. Ω προ το αν τελικά τα ευρωπαϊκά αυτά χρήματα δημιούργησαν μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Συντοπείτε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πραγματικό κίνδυνο εδώ. Και θα να συζητήσουμε τα ζητήματα αυτά και με τους νέους γεωργούς, οι οποίοι είναι πολλές φορές οι χαμένοι σε όλα αυτά τα καθεστώτα ευελιξίας. Ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Δευθυντή Κοτορούνη. Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να απαντήσω σε ένα από τα ερωτήματα που ετέθη σχετικά με τους νέους γεωργούς και ποιες είναι οι προθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε περισσότερα πράγματα από αυτό που επιτρέπεται να γίνει σε επίπεδο κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη μπορούν να ανακατανείμουν κάποιες πληρωμές και ένα 30% του εθνικού φακέλου του χρηματοτικού μπορεί να δοθεί σε τέτοια ανακατανομή που σημαίνει ότι μπορούν πόροι να μεταφερθούν από μεγάλες σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Αλλά είδαμε ότι ελάχιστα κράτη-μέλη τελικά χρησιμοποίησαν αυτή τη δυνατότητα. Και ας μην αναφερθώ και σε όλα τα υπόλοιπα εργαλεία τα οποία εφίστανται στα πλαίσια του συστήματος άμεσων ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητα, της πλήρου σύγκλησης ή της ε, μερικής τουλάχιστον σύγκλησης που εν μέρη τουλάχιστον θα διευθετούσε τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν για του νέου γεωργούς τα εργαλεία, τα μέσα υφίστανται. Το ζήτημα περισσότερο είναι κατά πόσο όντω τα χρησιμοποιούν ή αν τα χρησιμοποιούν ορθά τελικά τα κράτη-μέλη και αν όντω έχουν χρησιμοποιήσει σωστά την ευελιξία για να επωφεληθούν τελικά οι νέοι γεωργοί. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονε μα ήθελα να κάνω και εγώ λίγα σχόλια. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Γεωργία είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένη ε, λόγω μετεωρολογικών συνθήκων, διαφορετικούς τρόπους παραγωγής, διαφορετικά προβλήματα, άλλες παραδόσεις, διαφορετικά μεγέθη των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ορεινές και παιδινές περιοχές. Μεγάλη διαφοροποίηση. Γι' αυτό και χρειάζεται διαφοροποίηση και στην εφαρμογή της κοινή πολιτικής. Ε, αν δεν είναι προσοδοφόρια παραγωγή σε ορισμένες περιοχές, ε, ε θα εξαφανιστεί η γεωργία από τις περιοχές αυτές. Ταυτόχρονα θα πρέπει και να φροντίσουμε να επιβιώσουν οι γεωργοί μας, αλλά να ληφθούν υπόψη και οι κανόνες του ανταγωνισμού. Δεν θα πρέπει οι άμεσες ενισχύσεις να διαταράσουν τον θεμητό ανταγωνισμό ή να διαταράσουν την παραγωγή. Επίσης, αυτό σίγουρα επηρεάζει και τον τρόπο πληρωμής σε επίπεδο κράτους μέλους. Και αν ε, εφαρμόσουμε γενικότερα κάποιε διατάξει, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τι δημοσιονομικέ δυνατότητε που έχουν κάποια κράτη-μέλη να προβαίνουν σε μεγαλύτερε ε, πληρωμές. Επίση υπάρχει το θέμα τη πρόσληψης, τα οικονομικά προβλήματα, η εγκατάλειψη μερικέ φορέ κάποιων περιφερειών και περιοχών όπω μα είπε η κυρία Σένερα. Πώ θα τα λάβουμε και αυτά υπόψη στην κοινή γεωρική πολιτική ή στη χορήγηση ευελιξίας. Δέκα λεπτά το πολύ παρακαλώ, θα ξαναδώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας για να απαντήσουν. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας. Θα ήθελα να σταθώ σε μερικές από τις ερωτήσεις σας. Καταρχήν σας ευχαριστώ θερμά για τις πολύ εύστοχες ερωτήσεις και τα οξυντερική σας σχόλια. Σίγουρα η ευελιξία είναι ένα από τα θέματα της κοινή γεωργικής πολιτικής που πραγματικά αξίζει να συζητηθούν εκτενώς. Και πολλές ε, ερωτήσεις και σχόλια περιλάμβαναν κάποιες επιφυλάξεις και ανησυχίες για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει ευελιξία στον ε, ανταγωνισμό ή στην ικανότητα για ε, τη δυνατότητα υλοποίηση ε, των στόχων τη κοινή γεωργική πολιτική και κατά πόσο η ευελιξία συμβάλλει στην υλοποίηση αυτών των στόχων. Εγώ θεωρώ ότι η δημόσια πολιτική αρχίζει σε επίπεδο αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων πρώτα απ' όλα. Και όσο και να συζητάμε για τους στόχους ε, της κοινή ζωρικής πολιτικής σε γενικό και όριο ε, στο επίπεδο, δηλαδή βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, ε, αηφόρος, διαχείριση των φυσικών πόρων, ζωτικότητα και συνοχή των αγροτικών περιφερειών. Αυτά είναι εύκολο να τα συζητούμε στη θεωρία, αλλά όσο επισέρχεται κανείς στη λεπτομέρεια και ξεφεύγει από τις γενικότητες, προσκρούει σε δυσεπίλητα προβλήματα. Και εκεί θα πρέπει για να λυθούν αυτά τα προβλήματα να δοθούν κάποια ανταλλάγματα, να γίνουν κάποιες αντισταθμίσεις. Όπως το θέμα της ε, στρέβλωσης του ανταγωνισμού και των συνδεδεμένων ενισχύσεων. Θα πρέπει να υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί τις στοχευμένες ενισχύσεις για την αντιμετώπιση κάποιων ειδικών διαρθρωτικών προβλημάτων που αφορούν συγκεκριμένους τομείς παραγωγής. Και στο μέτρο που γίνεται αυτό, ε, το πρόβλημα διορθώνεται. Αν όμως υιοθετήσουμε διαφορετικό πρίσμα και σκοπιά, δηλαδή πέραν της ε, επίλυσης κάποιων διαρθρωτικών προβλημάτων και ε, δούμε την κατάσταση σε δύο παρόμοιες αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε γειτονικές χώρες με παρόμοιες συνθήκες παραγωγής αλλά με διαφορετικά καθεστώτα εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει στρέβλωση. Κανονικά και οι δύο αγροτικέ εκμεταλλεύσει θα πρέπει να λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο ενισχύσεων με βάση τα κριτήρια. Αλλά εξαιτία τη ευελιξία και τη διακριτική ευχαίρεια που παρέχουμε στα κράτη-μέλη, η τρόπο εφαρμογή τη πολιτική στι δύο περιπτώσει, παρόλο που είναι παρόμοιε, είναι διαφορετικό. Και άρα τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά και στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Κάτι τέτοιο είναι μια αναπόφευκτη συνέπεια αν, αν θέλουμε να, διασφαλίσουμε αυτό το επίπεδο στοχοθέτησης. Οπότε θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα των στόχων. Και αν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο στοχοθέτησης και τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν όλα τα διαρθρωτικά, κοινωνικο-δημογραφικά ή φυσικά προβλήματα μέσω της ΚΑΠ αναπόφευκτα θα προσκρούσουμε σε τέτοιου είδου δευτερεύοντα προβλήματα όπω είναι τη αδικία, το θέμα του ανταγωνισμού. Το ίδιο ισχύει και με το θέμα τη ιστορική αναφορά σε σχέση με το μέλλον έχουμε τι άμεσε ενισχύσει που καλύπτουν τι ιστορικέ ζημίε, με βάση τα ιστορικά δηλαδή κριτήρια αναφορά. και τώρα θέλουμε να είμαστε πιο διορατικοί και να λαμβάνουμε υπόψη το μέλλον σε ό,τι φορά τι άμεσε ενισχύσει και όχι το παρελθόν. Και εδώ ε, γίνεται ένα, δίνονται κάποια ανταλλάγματα, γίνεται μια αντιστάθμιση. Βλέπουμε περισσότερο το μέλλον παρά το παρελθόν. Όλα αυτά είναι περίπλοκα, αλλά είναι αναπόφευκτο να, ότι θα χρειαστούν κάποιες αντισταθμίσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει διεξοδική ανάλυση κατά πόσο ε, είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο και τι είδους αντισταθμίσεις πρέπει να δοθούν. Και αυτό είναι και το νόημα της δημόσιας πολιτικής, να εξετάσει λεπτομεριακά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ανταλλαγμάτων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που θα θέσει εκ των προτέρων. Το ίδιο ισχύει και με την αυξανόμενη περιπλοκότητα σε επίπεδο ταμείων σε ό,τι αφορά τους στόχους. Πολλοί από εσάς ζητήσατε ποσοτικοποιημένες αναλύσεις και αριθμητικά στοιχεία για τις συνέπειες της ευελιξίας στην πρόσβαση των νέων γεωργών. Δυστυχώς όμως η μελέτη μας ήταν πολύ οριθετημένη και είχε περιορισμένη εμβέλεια. Δεν μπορέσαμε να έχουμε πραγματικά διεξοδική ποιοτική ανάλυση της κατάστασης. Κάτι τέτοιο όμως μπορεί να γίνει με συνήθεις ε, έρευνες αξιολόγησης που θα περιλαμβάνουν και μια ποσοτικοποιημένη ανάλυση. Αυτά από μένα μπορεί η ίσως να συνεχίσει. Ευχαριστώ. Θα ζητώ συγγνώμη, ναι, τώρα άνοιξα το μικρόφωνο. Επί της ουσίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, η ευελιξία αποτελεί απάντηση στις διαφορετικές συνθήκες που υφίστανται από τη μία γεω... γεωργική δομή στην άλλη στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια γεωργικη δομη στην αλλη στα διαφορα κρατη μελη της ποικιλία και ένα υψηλό ποσοστό διαφορετικότητας. Αν θέλουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε όλα σε κεντρικό επίπεδο, σε ενωσιακό επίπεδο, αυτό θα ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα τελικά. Θα ήταν μάλλον αδύνατον να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τον ίδιο τρόπο μια κατάσταση στη Σλοβενία, στι κάτω χώρε, στην Ισπανία ή σε κάποια άλλη χώρα. Δεν μπορούμε να έχουμε μια ομοιόμορφη προσέγγιση παντού. Γι' αυτό το λόγο ευελιξία αποτελεί μια καλή λύση και μας επιτρέπει τελικά να αντιμετωπίσουμε τις πολλές και διαφορετικές συνθήκες που υφίστανται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από αυτό όμως, θα μπορούσε να προκύψει μια κατάσταση όπου οι γεωργοί καταλήγουν να την χάνουν διαφορετικής μεταχείρισης. Ένας γεωργός σε μια χώρα, για παράδειγμα, θα μπορούσε να λάβει μια επιδότηση για τον εξυγχρονισμό της εκμετάλλευσής του, ενώ ένας άλλος γεωργός σε μια άλλη χώρα μπορεί να έχει να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικές επιδοτήσεις. Εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει ένα συντονισμένο σύστημα και είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στους γεωργούς για ποιο λόγο ένας γεωργός στην Ολλανδία την χάνει συγκεκριμένη μεταχείριση ε, ή λαμβάνει επιδοτήσει τι οποίε δεν λαμβάνει ένα άλλο γεωργό στην Σλοβενία ή σε κάποια άλλη χώρα. Ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται χάρη στην ευελιξία είναι ότι η ευθύνη περνά από το νοσιακό στο εθνικό επίπεδο και να πόκειται τελικά στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν όπως αυτά κρίνουν ότι είναι καλύτερα τις πολιτικές της κοινή γεωργικής πολιτικής, ακριβώς επειδή υφίστανται εντελώ διαφορετικές συνθήκες και πολλές γεωγραφικές ιδιαιτερότητες. Είδατε έπειτα τα τρία διαφορετικά σενάρια προς την ευελιξία τα οποία σας παρουσιάσαμε. Και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το εφιστάμενο καθεστώς, δηλαδή η ευελιξία όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις και μη ευελιξία όσον αφορά τα μέτρα αγορά ότι αυτή ήταν τελικά η καλύτερη λύση. Ευελιξία όμως για τα μέτρα κοινή οργάνωση αγοράς. Θα μπορούσατε ουσιαστικά να μας ζητήσετε να έχουμε ευελιξία και για τα μέτρα αυτά. Πώς θα εφαρμοζόταν όμως μια τέτοια ευελιξία. Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα θα έπρεπε να μας απασχολήσει πρώτα. Και ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται και όλες αυτές οι συζητήσεις ε, για το Brexit. Και ουσιαστικά τίθεται και το ερώτημα ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια εθνική γεωργική αγορά και μια ενωσιακή κοινή αγορά. Αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται το θέμα αυτό, γιατί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάμε για μια κοινή μόνο αγορά γεωργικών προϊόντων. Τώρα, αν για τι άμεσε ενισχύσει δεν είχαμε την ευελιξία αυτή και είχαμε μια ομοιόμορφη προσέγγιση και εφαρμογή τους, πώς θα εφαρμοζόταν μια τέτοια προσέγγιση στην πράξη, θα ήταν δυνατή. Ακριβώς λοιπόν επειδή κάθε φορά προσπαθήσαμε να δοκιμάσουμε και το αντίθετο σενάριο, καταλήξαμε στο συμπέρασμα αυτό ότι το εφιστάμενο τελικά καθεστώς ευελιξίας αποτελεί όντως την καλύτερη επιλογή που έχουμε. Τόμας, θες να συνεχίσεις εσύ. Ναι, κάποιες ερωτήσεις υπάρχουν ακόμα. Ας πούμε η έλλειψη διαφάνειας και η περιπλοκότητα αναφερθήκαν ως κρίσιμα ζητήματα. Αυτό είναι αλήθεια. Αν δείτε τους κανονισμούς για την ευελιξία, είναι σχετικά κατανοητή. Αν όμως δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη με τους μεμονωμένους, μεμονωμένους γεωργούς και προσπαθήσετε να αποτιμήσετε τον αντίκτυπο της ευελιξίας στους νέους γεωργούς όπως επίσης να δείτε και τα γεωργικά προβλήματα και τα περιβαλλοντικά προβλήματα τότε ο βαθμός περιπλοκότητας αποτελεί πραγματικά βάρος για την αξιολόγηση και αυτό είναι η άλλη πλευρά, η άλλη μεριά του θέματος που δεν πρέπει να το ξεχνάμε όσον αφορά την ε, προσέγγισή μας. Μάλιστα. Ακούσαμε τις απαντήσεις των εμπειρογνωμόνων μας. Και σίγουρα η σημαντική και καρποφόρα ζήτηση που έγινε θα μας βοηθήσει και στο μέλλον για τη μεταρρύθμιση της γεωρικής πολιτικής. Ευχαριστούμε θερμά τους καλεσμένους μας για την ενδιαφέρουσα μελέτη που μας υπέβαλαν και που θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω ανάλυση και από εμά. Περνάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 4. Πρώτα απ' όλα όμως να καλωσορίσω στην αίθουσα τους επισκέπτες καλεσμένους από το Βαρδεβούργο της κυρίας Μέλχιορ. Καλώς ήρθατε. Καλή διαμονή στις Βρυξέλλες και καλώς ήρθατε και στη δική μας Επιτροπή της Γεωργίας. Περνάμε τώρα μετά τον χαιρετισμό των επισκεπτών στο επόμενο σημείο, το σημείο 4 όπως σας είπα. που αφορά την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου και ιδιαίτερα του κυρίου Βοητσεχόφσκι, του πρώην συναδέλφου και αντιπροέδρου της Επιτροπής Γεωργίας, τον οποίο και καλωσορίζω θερμά και πάλι στην Επιτροπή μας. κύριος Βοητσεκόφσκι είναι εξοικειωμένος με τους ε, κανόνες που ισχύουν στις συζητήσεις μας, δεν χρειάζεται να σε παραλάβω. Θα μας μιλήσει για το καθεστώς των νέων ε, γεωργών. Αναφέρθηκε και στην προηγούμενη συζήτηση η υποστήριξη για τους νέους γεωργούς και σίγουρα θα μας απασχολήσει και στο μέλλον αυτό το θέμα της στήριξης και της ενίσχυσης των νέων γεωργών, γιατί και στο μέλλον της ΚΑΠ θα έχουμε πρόβλημα με την, τη γύρεση του πληθυσμού στην Ήπεθρο, στις αγροτικές περιοχές και τι μέτρα και μηχανισμούς χρειαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε αυτή την ηλικιακή ανανέωση την ανανέωση των γενεών και να προσελκύσουμε όλο και περισσότερους νέους γεωργούς ε, στις αγροτικές δραστηριότητες. Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω στην εισαγωγή. Νομίζω πολύ καλύτερα θα το κάνει από μένα ο καλεσμένος μας ο κύριος Βοητσεχόφσκι σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Τσέσουαφ και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου έδωσαν να παρουσιάσω την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου που είναι η τρίτη έκθεση του Τμήματος Ελέγχου ένα ε, στο οποίο απασχολούμε ε, από τότε που ανέλαβα ως μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου και είναι και η πρώτη έκθεση που αφορά ακριβώς τους νέους γεωργούς, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φυσικά ευχαριστώ θερμά και την Επιτροπή Γεωργίας ε, για το ενδιαφέρον που δείχνει για αυτό το θέμα που θα είναι πολύ σημαντικό και για τις μελλοντικές συζητήσεις ε, για την κοινή γεωργική πολιτική. επιστρέφω λοιπόν εδώ μετά από ένα χρόνο και από τότε που ανέλαβα ως μέλος του ελεκτικού συνεδρίου. Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από το διορισμό μου. Χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι κοντά σας και θα ήθελα να πω ότι ελέγξαμε την ευρωπαϊκή στήριξη στους νέους γεωργούς και όπως λέει και ο τίτλος έκθεσης ε, αναφέρει το πρόβλημα που επισημάνουμε, δηλαδή ότι η μελλοντική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους νέους γεωργούς θα πρέπει να στοχοθετείται καλύτερα ώστε να συμβάλλει σε μια αποτελεσματική ε, ανανέωση των γενεών. Ποια είναι τα πιο ενδιαφέροντα πορίσματα καταρχήν της έκθεσής μας. Στην εισαγωγή της έκθεσης βρίσκουμε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Διαπιστώνουμε ότι ε, τελευταία δεκαετία μειώνεται ο αγροτικός πληθυσμός ο πληθυσμός των αγροτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005 μέχρι το 2013, δεν έχει περάσει καν δηλαδή ολόκληρη δεκαετία, σχεδόν μια δεκαετία, είχαμε μια μείωση του αγροτικού πληθυσμού από 14,5 εκατομμύρια το 2005 σε 10,7 εκατομμύρια το 2013. Έχει πάρει μια φθήνουσα πορεία λοιπόν ο αγροτικός πληθυσμός. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι Περίπου 4.000 μέσες αγροτικές εκμεταλλεύσεις τη δεκαετία το χρόνο χάνονται και περίπου 30.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις το μήνα χάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική πολιτική πρόκληση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε εσεί περισσότερο πολιτικοί και όχι εμεί ω ελεγκτέ. Θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση τη κατάσταση και να βρούμε τι κατάλληλε λύσει ώστε το μέλλον να αναχαιτήσουμε αυτή την απώλεια αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Και μάλιστα φαίνεται πώ μειώνεται ο αγροτικό πληθυσμό στα κράτη-μέλη ανά ηλικιακή ομάδα και σε κάθε ηλικιακή ομάδα έχουμε μείωση του πληθυσμού των γεωργών, των αγροτών και μάλιστα διαπιστώνουμε μείωση και του πληθυσμού των νέων γεωργών. Και μάλιστα στην ίδια περίοδο που εξετάζουμε, από το 2005 μέχρι το 2013, διαπιστώσαμε ότι μειώθηκε και ο ρυθμός των νέων γεωργών από 3,3 εκατομμύρια το 2005 σε 2,3 εκατομμύρια το 2013. Χάσαμε δηλαδή ένα εκατομμύριο νέους γεωργούς μέσα σε 8 χρόνια. Να σας δείξω και μια γραφική απεικόνηση που μας δείχνει παραστατικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Βλέπουμε σε αυτό το γράφημα τη μεσαία κόκκινη γραμμή που δείχνει τη συμμετοχή στον πληθυσμό των νέων γεωργών. Που όταν λέμε νέοι γεωργοί εννοούμε για στατιστικούς σκοπούς γεωργούς κάτω των 44 ετών. Αυτή στατιστικά είναι νέοι, θεωρούνται νέοι κάτω των 44. Και γενικώ στην κοινωνία το ποσοστό τους είναι περίπου 40%. Το 40% του πληθυσμού είναι κάτω των 44 ετών. Και το, η γαλάζια γραμμή αφορά την απασχόληση αυτής της ηλικιακής ομάδας που είναι περίπου 50% γενικώ και στην γεωργία μόνο το 20% των απασχολουμένων είναι νέοι. 20% δηλαδή των ε, γεωργών είναι κάτω των 44 ετών και 80% των γεωργών είναι άνω των 44 ετών. Εδώ έχουμε μια άλλη γραφική παράσταση που δείχνει τον πληθυσμό των αγροτών. Η χαμηλότερη γραμμή ε, δείχνει τη μείωση από 3,3 εκατομμύρια σε 2,3 εκατομμύρια μέσα σε 8 χρόνια και η κόκκινη γραμμή δείχνει το μέσο μέγεθος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που κατέχονται από νέους γεωργούς και που έχει αυξηθεί. Ήταν περίπου 12 εκτάρια ή μάλλον όχι λάθος λέει ο κύριος Βοτσεχόφσκι ε, Ήταν από 18 περίπου εκτάρια ο μέσος όρος αγροτικής εκμετάλλευσης των και έχει πάει ε, στα, 24. Έχει αυξηθεί το μέγεθος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που κατέχονται από νέους. Επίσης βλέπουμε ε, το 2005 57,7 εκατομμύρια εκτάρια σε νέους Γιώργους και 51,9 εκατομμύρια το 2013. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παράρτημα στην έκθεσή μας. Το παράρτημα υπαριθμών 2. Σας παραπέμπω στο παράρτημα 2 που περιλαμβάνει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που δείχνουν την κατάσταση ανακράτος μέλος. Αν δούμε την κατηγορία των νεότερων γεωργών, κάτω των 35 ετών δηλαδή, βλέπετε την αριστερή στήλη του πίνακα, μόνο σε δύο χώρες μέλη, μόνο σε δύο χώρες μέλη το ποσοστό των νέων γεωργών κάτω των 35 υπερβαίνει το 10%. Μόνο στην Αυστρία και στην Πολωνία έχουμε τέτοιο ποσοστό. Ενώ στην άλλη στήλη, η γεωργοί που είναι άνω των 65 ετών, η άκρα δεξιά στήλη του πίνακα, βλέπουμε ότι μόνο σε τρεις χώρες το ποσοστό των γεωργών άνω των 65 ετών έχουν ποσοστό κάτω του 10% ηλικιωμένων γεωργών. Δηλαδή στη Γερμανία, την Αυστρία και την Πολωνία έχουμε ηλικιωμένου γεωργού κάτω του 10% του συνολικού γεωργικού πληθυσμού. Ε, σε πολλά όμως κράτη-μέλη έχουμε μεγάλα ελύτερα ποσοστά ηλικιωμένων και μάλιστα στην Πορτογαλία πάνω από 50% των γεωργών είναι άνω των 65. Βλέπετε λοιπόν τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την ηλικιακή κατανομή των γεωργών. με έντονο πράσινο χρώμα βλέπετε τις χώρες στις οποίες λαμβάνει η χώρα κάποια ηλικιακή ανανέωση, κάποια ανανέωση των γενναιών γεωργών. Για παράδειγμα, αυξάνεται το ποσοστό των νέων γεωργών στη Βουλγαρία, για παράδειγμα και στις δύο κατηγορίες, και κάτω των 35 και κάτω των 44 έχουμε αύξηση των νέων γεωργών. Το ίδιο και στη Γερμανία. Στη Γαλλία είναι μικρή αύξηση στην πρώτη ηλικία και ομάδα, κάτω των 35. Στη Λιθουανία, Μάλτα και στη Ρουμανία και στις δύο κατηγορίες, ε, Σλοβενία και Σλοβακία το ίδιο. Και στη δεξιά στήλη έχουμε τα κράτη-μέλη στα οποία βλέπουμε μείωση του ποσοστού των ηλικιωμένων γεωργών, των, άνω των 65 δηλαδή ετών, στη Βουλγαρία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Λιθουανία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία έχουμε μείωση του ποσοστού των ηλικιωμένων γεωργών άνω των 65. Πάντως στην πλειοψηφία των κρατών μελών δεν διαπιστώνουμε σημαντική ηλικιακή ανανέωση. Δυστυχώς μειώνεται το ποσοστό ανανέωσης των γενεών στα περισσότερα κράτη-μέλη. Ποια είναι τα βασικά πορίσματα τώρα της ε, έκθεσης ε, του Ελεκτικού Συνεδρίου και ποια είναι, ε, ποιες είναι οι βασικές μας συστάσεις. Ah, sorry, <laughs> that is, yes. First I'd like to... Καταρχήν, να σας υπενθυμίσω ποιες ήταν οι ερωτήσεις που θέσαμε στον έλεγχο που πραγματοποίησαμε. Η ερώτηση ήταν, η, η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους νέους γεωργούς είναι καλά σχεδιασμένη ώστε να συμβάλλει σε ουσιαστική βελτίωση της ανανέωσης των γενναιών στη γεωργία. Αυτή ήταν η ερώτηση που θέσαμε προκειμένου να πραγματοποιήσουμε, να διενεργήσουμε αυτόν τον έλεγχο. Πού έγινε ο έλεγχος σε τέσσερις χώρες μέλη, στη Γαλλία, στην χώρα του Λίγυρα και στα Μιντή Πυρηναία, στην Ισπανία στην περιφέρεια της Ανταλουσίας, στην Πολωνία στη Βαρμία, Μαζουρία και στην Κάτω Σιλεσία και στην Ιταλία στις περιφέρειες της Εμιλίας Ρωμάνια και της Πούλιας. Ποια είναι τώρα τα βασικά συμπεράσματα, τα κύρια πορίσματα της έκθεσής μας. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι στόχοι της ε, κοινοτικής υποστήριξης δεν είναι καλά προσδιορισμένοι και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα και οι συνέπειές τους δεν είναι σαφή. Και ποιες, ε, ποια είναι η σύστασή μας μετά από τα συγκεκριμένα συμπεράσματα είναι ότι πρέπει να καθοριστεί, προσδιοριστεί καλύτερα ποιο θα πρέπει να τύχει υποστήριξη και ποια θα πρέπει να είναι τα αναμενόμενα ή τα προσδοκόμενα αποτελέσματα τη ευρωπαϊκή αυτή συνδρομή. Τα επόμενα συμπεράσματα οι ουσιαστικές ανάγκες, οι αυθεντικές ανάγκες των νέων γεωργών δεν αναλύθηκαν δεόντως και ως εκ τούτου η μορφή, το ποσοστό και το χρονοδιάγραμμα της ενίσχυσης μόνο μερικώς ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νέων γεωργών. Οπότε η σύστασή μας είναι να βελτιωθεί η λογική της παρέμβασης ενισχύοντας τη αξιολόγηση των αναγκών και ορίζοντας στόχους που θα είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι. Άλλο συμπέρασμα είναι ότι δεν ήταν σαφω στοχοθετημένα τα μέτρα τη στήριξη. Θα πρέπει να βελτιωθεί λοιπόν η στοχοθέτηση των μέτρων προκειμένου να εμφανιστούν οι νέοι γεωργοί να παραμείνουν στην Ήπεθρο. Και το τελευταίο αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε ελάχιστε αποδείξει ότι η ευρωπαϊκή στήριξη διευκόλυνε την εγκατάσταση των νέων γεωργών και βελτίωσε την ανανέωση των γενναίων. Οπότε η σύστασή μας είναι να βελτιωθεί η παρακολούθηση ε, και το σύστημα αξιολόγησης προκειμένου να συγκεντρωθούν τα κατάλληλα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πολιτικής μας. Κυρίες και κύριοι αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, αυτά ήταν εν ολίγη τα συμπεράσματα της έκθεσης του Ελεκτικού Συνεδρίου που καταδεικνύει ότι οι νέοι Γεωργοί αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα, αλλά δεν είναι οι μόνοι που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υπάρχει ένα πρόβλημα αποτελεσματικότητας τη κοινή γεωργική πολιτική που πλήττει όλες τις ε, ηλικιακές ομάδες των γεωργών και ελπίζω η έκθεσή μας να αποτελέσει τη βάση για μια διεξοδική και σημαντική συζήτηση για το μέλλον της κοινή γεωργικής μας πολιτικής και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Συγγνώμη, να σας ενημερώσω ότι μου κάθεται ο κύριος Λορέντζο Τιρέλη, που είναι ο επικεφαλής του κλιμακίου ελέγχου. Η κυρία ε, Καμόρους ε, είναι η ε, επικεφαλής του γραφείου μου και είναι και στη διάθεσή σας να απαντήσω σε απορίες σας και φυσικά και εγώ στο μέτρο που δίναμε. Ευχαριστώ κύριε Βοτσεχόφσκι. Περνάμε στη συζήτηση, ευχαριστώντας και πάλι θερμά τον κύριο Γιάννος Βοτσεχόφσκι για την παρουσίαση της αιτήσιας έκθεσης του Ελληνικού Συνεδρίου, της ειδικής έκθεσης του Ελληνικού Συνεδρίου και ευχαριστούμε φυσικά και τους συνεργάτες του. 1,5 λεπτό παρακαλώ καθένα. η κυρία Ράς Γκαρσία πρώτη. Κύριε Βοτσεχόφσκι, ευχαριστώ. Είστε γνωστός εδώ της Επιτροπής μας και με χαρά σας ακούσαμε. Κάπως εξεπλάγει από αυτά που είπατε και συμμερίζομαι την άποψη τη δική σας ότι η αλλαγή, η ανανέωση το γυρών είναι σημαντική, αλλά τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Εμείς στη χώρα μου θεωρούμε ότι το 3% των ε, γεωργών είναι 135, τώρα είναι 0,7. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα φοβερό, πάνε σχετικά καλά τα πράγματα στην Ισπανία. Αλλά νομίζω μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Ήδη είπε η Ισπανία στο Συμβούλιο Είπε λοιπόν ότι μια σημαντική θέση θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε τον κανονισμό Omnibus για να ρυθμίσουμε αυτά τα θέματα που δεν πάνε καλά. Οπότε εντάξει αυτά τα μέτρα, αλλά να είναι συγκρίσιμα ο πρώτος και ο δεύτερος πυλώνας. Εσείς επικρίνετε ας πούμε την Ανταλουσία και λέτε διάφορα ότι καταρχάς η περίοδος είναι πολύ μακροσκυλής για την ε, ρυθμίση των εκκρεμωτήτων. Αλλά η άμεσα προηγούμενη περίοδος είναι εξίσου κακή με το 2005-2007. Να σας υπενθυμίσω ότι τότε στην Ανταλουσία είχαμε 17 μήνες μέχρι το 2013. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε τώρα, από το 2014 και μετά, να μου το διευκρινίσετε. Μετά, είναι αλήθεια ότι η Ανταλουσία δαπάνησε τα χρήματά στο 2015 και το 2016, οπότε εφ' δεν έχει χρηματικούς πόρους για να βρει λύσεις. Όμως ρωτάω, θα μπορούσε η ανταλουσιανή κοινότητα να μεταβιβάσει πόρους από την ανάπτυξη της υπέθρου για να βοηθήσει αυτούς τους νέους γεωργούς που είναι τόσο ε, σημαντικοί. Αυτά. Και αν έχετε βρει και κάποιο άλλο σφάλμα για την κοινότητα της Ανταλουσίας, να μας το πείτε. Αλλά αυτά είναι και χρήσιμα και απαραίτητα και θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Κύριος Καπούτο. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Βασεκόφσκι για την έκθεσή του και το συνεργάτης του που ως έκθεση θεωρώ πολύ χρήσιμη. Και εγώ είμαι και εγώ συνεισηγητής για τα προγράμματα που αφορούν τους νέους γεωργούς. Συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν για το ότι βασιζόμαστε σε μια λογική που δεν είναι σαφώ προσδιορισμένη και νομίζω είναι και ακατάλληλη. Δεν προσδιορίζει λοιπόν τα αποτελέσματα και τα προσδοκόμενα ωφέλη. Θα πρέπει λοιπόν για να προωθήσουμε την ανανέωση των γενεών να κάνουμε κάτι πιο στοχευμένο. Όσον αφορά τώρα τις ενισχύσεις για τους νέους γεωργούς, και εγώ βλέπω να μην υπάρχει συντονισμό του πρώτου πυλώνα και των μέτρων εκεί με το δεύτερο πυλώνα, ούτε και με τα εθνικά, με τους πυλώνες. Για την εποπτεία επίσης. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Επειδή ακριβώς δεν έχουμε σοβαρούς δείκτες εδώ, δηλαδή οι χρήσιμους δείκτες, ώστε να κατανοήσουμε πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε αυτή την αξιολόγηση που κάνουμε. Βεβαίω θα πρέπει να βελτιώσουμε και τη λογική της παρέμβασης, ε, αποτιμώντας τις ανάγκες, τους στόχους, σε σχέση με τον γενικότερο στόχο, δηλαδή της πρόθεσης της ανανέωσης των γενναιών. Επίσης θα πρέπει να έχουμε πιο στοχευμένα μέτρα, τα οποία αποβλέπουν ακριβώς την επιλογή των προγραμμάτων, χρησιμοποιώντα επίσης και σχέδια επιχειρηματικά. Θα έχουμε την ευκαιρία στο μέσο μέλλον να συζητήσουμε περισσότερο σε βάθος αυτά τα ζητήματα και υπενθυμίζω ότι ζητήθηκε η μελέτη από την Κομάγκρη η οποία θα συζητηθεί προσεχώς στο Κοινοβούλιο ώστε να έχουμε την ευκαιρία, θα ήταν καλό αυτό να γίνει, ώστε να έχουμε την ευκαιρία να συγκρίνουμε ακριβώς αυτές τις δύο εκθέσεις. Ευχαριστώ. Ναι, όντω είστε ιδιαίτερα εξοικειωμένο με το θέμα αυτό. Ναι, και έχετε αναλάβει το σχετικό πόνημα. Αλλά ο χρόνος πιέζει. Παρακαλώ, κύριος Λαζό. Oui, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, αν θέλουμε να υπάρξει ένα νέο των γενεών, θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε πολλά να κάνουμε. Και το πρώτο μέτρο θα ήταν βέβαια να σταματήσουμε τις πολιτικές που υπάρχουν και που τις βλάπτουν. Να υπενθυμίσω ότι είχαμε 14,5 εκατομμύρια γεωργού το 5, 10, το 13, λιγότερου από δεν ξέρω πόσα σήμερα. Βλέπετε λοιπόν ακριβώ την μείωση, το φθήνοντα αριθμό. Αυτό που ε, αποθαρρύνει σήμερα είναι οι συνθήκε εργασίας, οι δύσκολε, όπως ξέρετε, αλλά και το γεγονό ότι τα εισοδήματα αυτά δεν επαρκούν. Υπάρχουν προβλήματα με χρέη κλπ. Και εγώ ο ίδιος δεν έχω σε ποιους να παραδώσω τη δραστηριότητά μου. Εμείς δεν θέλουμε μόνο ενισχύσεις, αλλά σωστές τιμές. Τώρα για τα υπόλοιπα που συζητάμε, επειδή είμαι και περιφερειακό σύμβουλο από το 4, ε, να πω ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, ιατρική κάλυψη, περίθαψη κτλ. Ε, όλα αυτά δεν έχουν βελτιωθεί. Οπότε είναι δύσκολο να ενθαρρύνει κανεί του νέου γεωργού να εγκατασταθούν σε κάποιε περιοχέ. Οπότε θα πρέπει να του ακούσουμε και του ίδιου. Θα πρέπει να του ακούσουμε αντί να του επιβάλλουμε έντρα χωρί να του ακούμε. Επίση, διαπιστώνω ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού μεταξύ χωρών μελών και ένωση Κάποιοι νέοι θεωρούνται, θε, θεωρείται ότι λαμβάνουν υπερβολικές ενισχύσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε ακριβώς την πίεση προς τις χώρες μέλη ακριβώς. Μήπως εξάλλου αυτό θα πρέπει να ήταν και στόχος της έκθεσης. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους εισηγητές για αυτή την έκθεση, την πολύ ενημερωτική αλλά και ενσυχητική. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς, αν υπάρχει ηλικιακό όριο για την παροχή της ενίσχυσης, αυτό δεν μας βοηθάει και πολύ. Δηλαδή, αν έχουμε ένα όριο 45 ετών, ας πούμε, θα πρέπει η ενίσχυση να δίνεται και σε αυτούς που είναι πιο νέοι. Επίσης, θα πρέπει να βοηθάμε τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες χρειάζονται βοήθεια και να ενισχύσουμε τις οικογένειες που δουλεύουν εκεί. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τις ε, επιχειρήσεις. Ακούστε, να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή, μήπω θα μπορούσαμε να του βοηθήσουμε από την αρχή, να δούμε ακριβώ τι άλλε δυνατότητε υπάρχουν, ώστε να του βοηθήσουμε και να του ε, κρατήσουμε στην γεωργία και να του ε, επιτρέψουμε να κάνουν τη δουλειά του. Όσοι αναλαμβάνουν ε, την επιχείρηση θα πρέπει να βοηθηθούν. Οπότε αυτό θα πρέπει να το πούμε εδώ ξεκάθαρα. Δεν θα πρέπει να το αναφέρουμε απλά και μα. Θα πρέπει να το τονίζουμε. Ναι, πρώτα ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Σικώσκη για την ε, έκθεσή του και την παρουσία του. Πράγματι, για το θέμα των γενεών αυτό είναι θέμα πολύ σημαντικό. Τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά. Είναι και ενδιαφέρουσα η έκθεση από αυτού. Βεβαίω, θα μπορούσαμε να συστήσουμε μια ε, καλύτερη παρακολούθηση στο στοιχείων που αφορούν τους νέους γεωργούς για να δούμε πώς εξελίσσονται. Αλλά νομίζω ότι λείπουν κάποια στοιχεία ποιοτικά. Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε σωστές επιλογές ε, για την ε, μελλοντική μεταρρύθμιση για τους νέους. Να δούμε ακριβώς τι γίνεται με τα στοιχεία ας πούμε, για τις εκμεταλλεύσεις, για τις εγκαταστάσεις, μετά πώς εξελίσσονται κάποια χρόνια μετά από την έναρξη της λειτουργίας τους. Θα δούμε ακριβώς λοιπόν τι ποσοστό, σε τι ποσοστό είναι επιτυχής αυτές οι ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις. Να δούμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε και τους λόγους αποτυχίας. Ε, στοιχεία λοιπόν και δεδομένα ποιοτικά ώστε να βαθύνουμε στι αξιολογήσει μα. να δούμε ακριβώς ποια είναι τα αίτια τη αποτυχία, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε κάποια στοιχεία απάντηση στι μελλοντικέ μεταρρυθμίσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχαμε δεχθεί πιέσει στην προηγούμενη θητεία από νέου ε, γεωργού λέγοντα ότι θα πρέπει να βοηθήσει η Επιτροπή του νέου ε, γεωργού, αλλά στην ουσία αυτό ήταν αδύνατο. Και η Κομισιόν ε, είχε αυτή την ιδέα το να αυξήσει ακριβώ τι πληρωμέ σε κάποιε περιοχέ για του νέου. Αλλά στην ουσία αυτά είναι πρόχειρα πράγματα, μπαλώματα. Και απλά και μόνο δώσαν περισσότερα χρήματα αυτή η Νέα Γεωργία και τίποτα άλλο. Είναι δύσκολο λοιπόν να λέξει κανεί μια παρόμοια κατάσταση. Και νομίζω ότι πραγματικά εδώ ακολουθούμε τελείω ασφαλμένο δρόμο. Αυτό ο όρο ανανέωση γενεών έχει γίνει έτσι ένα σύνθημα πια. Και θα πρέπει όμως να δούμε πού βρίσκεται το πρόβλημα, γιατί στη χώρα μου οι καλές γεές φαίνεται να εκμεταλλεύονται από κάποιους που δεν ξέρω κατά πόσο αφορά η κρίση, αλλά να σας πω επίσης ότι η κατάσταση ας πούμε στην Ουαλία και ήταν και σε ένα έντυπο πρόσφατα αυτό, αυτή η υπόθεση ο ένας κτηνοτρόφος μπόρεσε να αγοράσει ένα μερίδιο της επιχείρησης και μετά προσέγγισε και άλλους γεωργούς ακολουθώντας το ίδιο μοντέλο επειδή ακριβώς ε, έτσι είχε ενισχύσει τη φήμη του και μπόρεσε να εμπλέξει και άλλους νέους ε, γεωργούς ως υπεργολάβους, κάτι το οποίο θεωρώ ήταν ε, πολύ αξιόλογος τρόπος και λύση. Ήξερε λοιπόν τι έκανε και θα ήθελα να έρθει αυτός ο νέος εδώ, σε αυτή εδώ την Επιτροπή εδώ, να σας πει περισσότερα. Ευχαριστώ κύριε Αγγιλέρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο κύριος Βασικόσκη να τον καλωσορίσω και μας παρουσιάσει μια τόσο σημαντική έκθεση. αναφέρθηκε σε ανησυχητικά συμπεράσματα εκ μέρους του Ολεκτικού Συνεδρίου. Ε, είπαμε ότι για τους νέους οι στόχοι της ΚΑΠ δεν έχουν οριστεί σωστά. Επίσης οι ανάγκες των νέων δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Η στήριξη προς αυτούς δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αυτά είναι δηλώσεις που πραγματικά μας δείχνουν ότι κάτι συμβαίνει εδώ σε σχέση με τους νέους παρά τα μέτρα που έχουμε λάβει. Κάτι πάει καλά. Μια συγκεκριμένη ερώτηση να κάνω. Εδώ είδαμε ότι η τωρινή μεταρρύθμιση έγινε με την ε, συμβολή το 2% για τι άμεσε ενισχύσει για του νέου. Οι χώρε μέλη λένε ότι δεν μπορούν να δαπανίσουν αυτά τα χρήματα, κάτι το οποίο είναι ανήκουστο. Ανήκουστο. Μήπως θα πρέπει κάτι να αλλάξουμε λοιπόν για αυτό το 2%. Πάντως να σας ρωτήσω εγώ το εξής. Για την Ισπανία εμπειρία την ε, συναδελφό μου την κυρία Εράν ότι η Ισπανία τα πάνε καλά εκτός από την Ανταλουσία, δηλαδή την δικιά μου την περιφέρεια, που έχει το 25% της τελικής γεωργικής παραγωγής της χώρας ολόκληρης και που διαχειρίζεται όσο καμία άλλη τους πόρους αυτούς. Θα ήθελα λοιπόν να μου πει, όχι συγκεκριμένα, αλλά για ποιο λόγο θεωρεί ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα εκ μέρου του κράτους να ασκήσει αποτελεσματική πολιτική ώστε δηλαδή να υπάρξει κατάλληλη ενσωμάτωση των νέων στο κλάδο της Γεωργίας. Βλέπουμε ότι έχουμε αυτό το ποσοστό νέο το οποίο είναι χαμηλό. Είπαμε ότι δεν υπάρχει ανανέωση. Οπότε ε, ποιο είναι το μεγάλο εμπόδιο εδώ. Ευχαριστώ. Ο Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Βασικόφσκι, νομίζω ότι οι πληροφορίες μας δώσατε είναι πολύ ενδιαφέρουσες, μας αφορούν άμεσα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Μας δείξατε μια πολύ ενδιαφέρουσα γραφική παράσταση, ένα πίνακα μάλλον, με διαφορετική κατάσταση που ισχύει σε κάθε κράτος μέλος. Εξτάστε καθόλου τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας στα κράτη αυτά. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, που είπατε ότι έχουμε θετικά παραδείγματα. Είπατε ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας εκεί λειτουργούν θετικά υπέρ των γεωργών οι οποίοι μπορούν εύκολα να συνταξιδοτηθούν μετά την ηλικία των 60 ετών και μπορούν πολύ εύκολα να διαβιβάσουν στη συνέχεια την εκμεταλλευσή του σε κάποιον άλλον. Και μας είπατε έπειτα ότι για κάποιες άλλες χώρες τα πράγματα δεν είναι τόσο θετικά. Μήπως θα μπορούσαμε στο μέλλον να ασχοληθούμε και λίγο περισσότερο με τα συστήματα κοινωνική πρόνοιας τα οποία υπάρχουν στα κράτη-μέλη όσον αφορά τις πληρωμές των πρώτο πυλώνα θα πρέπει στα πλαίσια των ενισχύσεων αυτών να δούμε και τι γίνεται με τους συνταξιούχους ε, γεωργούς. Νομίζω ότι και αυτή την πτυχή θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας για το μέλλον. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά τον ορισμό του νέου Γεωργού, θέλω εδώ μία λογική εξήγηση, γιατί την έχουμε ζητήσει εμείς από τη Ρουμανία και νομίζω ότι το πρόβλημα αυτό υφίσταται και έχει εντοπιστεί και σε άλλα κράτη-μέλη. πρέπει να τεθούν κάποιες νέες προϋποθέσεις πέρα από την προϋπόθεση της ηλικία. Λέμε ότι ο γεωργός θα πρέπει να είναι ήδη ενεργό σε μια εκμετάλλευση. Ας πούμε ότι έχουμε όμως έναν Γεωργό, ο οποίο ηλικία 18 ετών είχε επενδύσει σε μια γεωργική εκμετάλλευση, πήρε μάλιστα και δάνειο από την τράπεζα, και τώρα είναι πια 25 ετών και χρειάζεται και περισσότερα χρήματα, και θέλει να κάνει μια αίτηση για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς, το Γεωργό αυτό, δεν του δίνουμε χρήματα. Νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα λογικό κενό το οποίο πρέπει να καλύψουμε. Δεύτερον, πολύ ωραίο το ότι επενδύουμε κοινοτικά κονδύλια για να βοηθήσουμε τους νέους γεωργούς να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της γεωργίας. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε και σε βάθος χρόνου να παρακολουθούμε τη δράση τους πολύ καλό να δίνουμε κονδύλια στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, αλλά όταν ξαφνικά σταματά το πρόγραμμα αυτό, τι κάνουμε. Εμείς θέλουμε να έχουμε βιώσιμες θέσεις απασχόλησης σε βάθος χρόνου και όχι να εξαφανίζονται οι θέσεις αυτές απασχόλησης μετά από 5-6 χρόνια. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τρόπον την να, να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Διότι αν τελικά χάνουν τη δουλειά τους, χάνουμε και εμείς χρήματα από την άλλη. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Βοσικόφσκι, τον ε, πρώην συναδελφό μας, για την εξαιρετική αυτή παρουσίαση. Ξέρετε ότι είχαμε συνεργαστεί για πάρα πολλά χρόνια. Ακούσαμε στην παρουσίασή σας ε, τις πολλές διαφορετικές συνθήκες που υφίστανται για τους νέους γεωργούς και οι οποίες ε, διαφοροποιούνται πάρα πολύ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Σίγουρα δεν θα πρέπει εδώ πέρα να επινοήσουμε εκ νέου τον τροχό. Ίσως θα πρέπει να κοιτάξουμε τα θετικά μοντέλα όπως αυτό της Αυστρίας, όπου οι νέοι γεωργοί καταβάλουν χαμηλότερες συνεισφορές κοινωνικής ασφάλισης από ό,τι για παράδειγμα στη Γερμανία. ή βλέπουμε έπειτα διαφορετικές συνθήκες που ισχύουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο όσον αφορά την συνταξιοδότηση των γεωργών. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να δούμε και την πρόοδο της τεχνολογίας και πώς μπορεί αυτή να βοηθήσει την κατάσταση των νέων γεωργών. Ξέρετε ότι χάρη στις νέες τεχνολογίες μπορεί κανείς να καλλιεργήσει πολύ πιο γρήγορα μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Στην ε, Βαβαρία, για παράδειγμα, έχουμε πολλούς νέους γεωργούς οι οποίοι ε, είναι ιδιοκτήτες ή εργάζονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Μήπως θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε περισσότερο στο ζήτημα των επενδύσεων. Μία γεωργική εκμετάλλευση 50 εκταρίων που λειτουργεί εύρυθμα, η οποία έχει ένα γόνιμο έδαφος. Αν συγκρίνεται μια τέτοια εκμετάλλευση με μια άλλη εκμετάλλευση των 50 εκταρίων που όμω το έδαφο δεν είναι σε καλή κατάσταση, τότε θα πρέπει στη δεύτερη προφανώ περίπτωση να κάνουμε πιο σημαντικέ επενδύσει. Ο κύριο Φλάναγκαν, ευχαριστούμε κύριε Βετζεχόφσκι για την έκθεση. Μπράβο Ε, ρωτήσατε αν ευρωπαϊκή στήριξη είναι καλά σχεδιασμένη και αν συμβάλλει στην ηλικιακή ανανέωση και καταλήξα στο συμπέρασμα ότι δεν επιτελεί του στόχους του αυτή η στήριξη. Και πολύ συχνά στην εκλογική μου περιφέρεια το διαπιστώνω ότι είναι υπερβολικά περιοριστικό το νέο σύστημα και έχει μία πενταετία σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των νέων γεωργών. Αυτή η προθεσμία δεν λαμβάνει υπόψη την περιπλοκότητα και την κυρίως της μεταβίβασης ή της ιδιοκτησίας α, ε, της γης και πολλοί νέοι γεωργοί ε, συμβάλλουν με διαφορετικούς τρόπους και τη στιγμή μπορούν να αναλάβουν οι ίδιοι την ε, εκμετάλλευση λόγω του, του περιορισμού του καθεστώτος ε, δεν μπορούν να τέχουν τις ενίσχυσεις γιατί τους λένε ότι έχετε ασχοληθεί με αυτό πάνω από μία πενταετία. Οπότε θα πρέπει να βελτιώσουμε αυτή την πρόταση. Ελπίζω να λύσουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται. Πάντως, σε τελική ανάλυση, ό,τι στήριξη και αν προβλέψουμε, αν οι γεωργοί δεν μπορούν να, να λάβουν μια καλή τιμή για τα προϊόντα τους. Αν δεν είναι βέβαιοι ότι θα έχουν διεξόδου στην αγορά, τότε δεν θα μπορέσουν ε, να εξασφαλίσουν το βιοπορισμό τους με τη Γεωργία. Πολλά πρέπει να αλλάξουν, αλλά είναι κρίμα όταν στην Ιρλανδία έχουμε... Ε, είχαμε μια, ένα φεστιβάλ για τη Γεωργία, διαπιστώνουμε ότι έχουμε περισσότερους ε, ε, γεωργούς κάτω των 35 από ότι ηλικιωμένους ε, γεωργούς άνω των 80. Σιγά μην ε, θριαμβολογήσουμε και όλα για αυτό το επίτευγμα. Ευχαριστώ κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Βοτσεχόφσκι για την παρουσίαση της ειδική έκθεσης. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα και σίγουρα θα πρέπει να βρούμε λύσεις ε, που θα προσανατολίζονται στο μέλλον και θα εξασφαλίζουν ε, βελτίωση της κατάστασης. Εμείς είχαμε αύξηση του αριθμού των γεωργών και των νέων. Έχετε όμως κάποια στοιχεία για τις αρρώσιμες, ε, τις επιφάνειες αρρώσιμων καλλιεργιών. Αυτές αυξήθηκαν ή μειώθηκαν. Γιατί ξέρω ότι οι αρρώσιμες καλλιέργειες, οι αρρώσιμες εκτάσεις αυξάνονται κάθε χρόνο ενώ είπατε ότι ο αγροτικός πληθυσμός ε, μειώνεται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυξάνεται η υποστήριξη αλλά στις μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ε, μια και όλο και περισσότεροι γεωργία καταλήγουν τη δραστηριότητά τους. Επίσης, οι νέοι γεωργοί και σε μας έχουν πρόβλημα με την ε, αγορά ε, της γης. Είναι πολύ δαπανηρή η αγορά της γης. Και επίσης είναι πολύ περίπλοκο το σύστημα. Ένας νέος γεωργός μπορεί να υπογράψει μια σύμβαση αγοράς, αλλά στην ουσία πρόκειται για μίσθωση. Και υπάρχει πρόβλημα ακόμη και στην ε, υπογραφή των συμβολέων πολλές φορές. Ο κύριος Κούσμικο, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τον ε, κύριο Βοτσεχόφσκι τον, το μέλος του ελεκτικού συνεδρίου και να τον συγχαρώ για την άρτια έκθεση που μας ε, υπέβαλε. Διαπιστώνουμε στην έκθεση σχετικά αρνητικές στάσεις ό,τι αφορά τους νέους γεωργούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε μία σχεδόν δεκαετία μειώθηκε ε, κατά 900.000 περίπου, αν δεν κάνω λάθος, ο αριθμός των νέων γεωργών. Χάσαμε σχεδόν ένα εκατομμύριο νέους γεωργούς μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία. Και στα κράτη-μέλη ή παρά τις μορφές συνδρομής που είχαμε για τους νέους γεωργούς, δεν καταφέραμε να στηρίξουμε τους γεωργούς κάτω των 44 ετών. Βέβαια, ε, είναι θετικό και πιο αισιόδοξο ότι στις νέες χώρες έχουμε καλύτερη ηλικιακή ανανέωση. Σε αντίθεση με τις παλιές 10 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η κατάσταση είναι πιο αρνητική. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών μελών. Εσείς πώς μπορείτε στο μέλλον, πώς πιστεύετε μπορούμε στο μέλλον να αξιολογήσουμε την ε, δαπάνη των κονδυλίων ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε την αποδοτικότητα των γεωργικών κονδυλίων στην κοινή γεωργική πολιτική κατά τη γνώμη σας και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόγκοβιτς Πολύ σημαντική έκθεση. Σας ευχαριστώ θερμά και τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Καταρχήν, γιατί οι νέοι Γεωργοί αποφασίζουν να μείνουν στο, στην οικογένειά τους και να αναλάβουν την οικογενειακή επιχείρηση. Γιατί θα το κάνουν, θα το κάνουν μόνο εφόσον μπορούν να επιβιώσουν, εφόσον μπορούν με την ανάληψη της οικογενειακής εκμετάλλευσης να εξασφαλίσουν το προστοζήν. Στα 65 δεν μπορεί κανείς να ανακυκλωθεί σε άλλο επάγγελμα, αλλά ο νέος μπορεί να λάβει την απόφαση, θα κρίνει. Αν είναι προσοδοφόρα και ελκυστική η γεωργική εκμετάλλευση, θα τη συνεχίσει. Αλλιώς θα κοιτάξει κάτι διαφορετικό να βρει. Μιλήσατε για την επιτυχία της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αυτή δεν θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των γεωργών. Η επιτυχία της ΚΑΠ θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι γεωργοί αυτοί έχουν ποιοτική ζωή, αν παράγουν ποιοτικά τρόφιμα, αν έχουν αξιοπρεπέ εισόδημα και ξέρουμε ότι η πλειοψηφία των ε, Ευρωπαίων Γεωργών είναι μικροκαλλιεργητέ. Τι να βγάλει κανεί σε 10-15 εκτάρια. Είναι πολύ μικρές οι καλλιέργειες αυτές, πολύ μικρές οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Και μειώνεται ο αριθμός των γεωργών, αλλά αυτό που προέχει είναι να τους δώσουμε τα εφόδια ώστε ε, να είναι προσοδοφόρα και βιοπεριστική η δραστηριότητά τους. Ήμουν κάποτε και υπουργό ε, Γεωργία στη Σλοβενία και χαίρομαι που είμαστε στην πράσινη ζώνη. Ε, στη Σλοβενία ε, έχουμε 5% των ενεργών γεωργών που είναι νέοι. Αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να καταπετρίσουμε σήμερα όλα τα αποτελέσματα, αλλά στο μέλλον θα είμαστε ικανοί να το κάνουμε. Οπότε για μένα τα συμπεράσματα είναι δύο. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους νέους γεωργούς ε, να έχουν πρόσβαση και σε μεγαλύτερες ε, γεωργικές εκμεταλλεύσει και να τους βοηθήσουμε να επιβιώσουν και επίση ποια είναι η κοινωνική κατάσταση των γονιών. Αν οι γονείς δεν έχουν καλή κοινωνική κατάσταση δεν θα ε, δώσουν κίνητρα στα παιδιά να αναλάβουν την οικογενειακή επιχείρηση. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους να ενθαρρύνουμε τους νέους να αναλάβουν γεωργική εκμετάλλευση και επίσης και τους ηλικιωμένους να μεταβιβάζουν την δική τους ε, γεωργική επιχείρηση. Ευχαριστώ. Δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε εδώ στην ανάλυση του προβλήματος των νέων. Γιατί κάποιος που είναι 45 ετών μπορεί να μην είναι νέος, αλλά είναι νέος γεωργός, δηλαδή ε, πρώτη εγκατάσταση στη γεωργία. Γιατί να μην ενθαρρύνουμε και αυτούς τους ε, γεωργούς. Το θέμα δεν είναι να ενθαρρύνουμε την ανασχόληση με τις γεωργικές δραστηριότητες μόνο και μόνο για την πρόσβαση στη στραματική ενίσχυση. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα ε, για την εγκατάσταση των νέων γεωργών με κάποια διάρκεια όμως, όχι ευκαιριακά. Επίσης, να εξασφαλίσουμε πρόσβαση των ε, νέων γεωργών και στην γεωκτησία στην πατρίδα μου είναι τόσο αστρονομικές ε, οι τιμές ε, των ακινήτων που δεν μπορεί, ο νέος δεν έχει πρόσβαση ε, στην ιδιοκτησία, στη ιδιοκτησία. Επίσης, πρόσβαση στο κεφάλαιο, στο δανεισμό. Δεν είναι όλες οι τράπεζες διατεθειμένες να δανείσουν σε νέους γεωργούς, γιατί θεωρούν τη γεωργία ρηψοκίνδυνη δραστηριότητα. Οπότε δεν χορηγούν εύκολα δάνεια. Επίση, πρέπει να φροντίσουμε ώστε και οι νέοι και οι λιγότερο νέοι να παραμένουν στην Ήπεθρο και να εξασφαλιστούν καλέ συνθήκε ε, για την αγροτική ανάπτυξη. Δηλαδή, η Ήπεθρό μα θα περιμωθεί και δεν θα μείνει κανένα πια στα χωριά. Θα εξαφανιστεί ο κοινωνικό ιστό. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε και στην αγροτική ανάπτυξη και όχι απλώς να μεταβάζουμε κονδύλια από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα. Ευχαριστώ. Κυρία Σένερα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω τρία σχόλια. Πιστεύω καταρχήν ότι η έκθεση που μας παρουσίασε πρόσωπος του Ελεκτικού Συνεδρίου είναι πολύ σημαντική και επιβεβαιώνει στην ουσία αυτό που διαπιστώνουμε και εμείς οι διεισόμαστε στις ε, περιφέρειές μας. Όλοι όσοι μένουμε στην Ήπεθρο βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πολλοί νέοι γεωργοί, δεν έχουμε εγκατάσταση νέων γεωργών όσο θα το επιθυμούσαμε. Ένα άλλο πρόβλημα έγκυται στο ότι η στήριξη για την εγκατάσταση των γεωργών δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες της νεολαίας. Η στήριξη προ, προορίζεται στην ε, ε, ενίσχυση των μεγάλων επενδύσεων. Αυτό τους ενδιαφέρει. Επίσης αναζητείται συγκεκριμένος οικονομικός στόχος για την εγκατάσταση. Απαιτούνται υπερβολικές επενδύσεις, κάτι που δεν δύναται να κάνει ο νέος και μερικές φορές ακόμη και τέτοια μεγαλεπίβολα επενδυτικά σχέδια αποτυχαίνουν. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι η ίδια η ΚΑΠ είναι αντικίνητρο για τους νέους Γιώργους, γιατί από τη μια δίνει ενισχύσεις και από την άλλη με την απορρίθμιση της παραγωγής, την απορρίθμιση των αγορών έχουμε κατακόρυφη πτώση των τιμών με αποτέλεσμα να μην είναι προσοδοφόρα η γεωργική δραστηριότητα. Δεν υπάρχουν προοπτικές για, μια, για έναν αξιοπρεπή βιοπορισμό από τη γεωργική δραστηριότητα. Άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η πρόσβαση στην αγορά της γη. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και επίσης σημαντικό είναι να διαφυλάξουμε και να θωρακίσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες στην Ήπεθρο. Τόσο στην παιδεία, την υγεία, αλλά και ε, τις δημόσιες υπηρεσίες ε, ε, παροχή συμβουλών για τις γεωργικές δραστηριότητες και υποστήριξη των αγροτών. Θα έδινα λοιπόν έμφαση σε αυτό το θέμα ώστε να καταργήσουμε το κριτήριο του συγκεκριμένου εισοδήματος από το επιχειρηματικό σχέδιο, γιατί ουσιαστικά αφορά κάποιου θεωρητικού υπολογισμού και δεν, δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα στη γεωργική εκμετάλλευση. Ευχαριστώ κύριο Σκαλινόφσκι. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον ελεγκτή μα. Οι δείκτε για την ανανέωση των γενεών στη Γεωργία, στα κράτη-μέλη, είναι πολλοί και διάφοροι και καταδεικνύουν και τεράστιες διαφορές σε ό,τι αφορά την ηλικιακή ανανέωση στη Γεωργία μεταξύ των κρατών μελών. Ακούσαμε προηγουμένως κάποια μελέτη για τη χορήγηση ευελιξίας ό,τι αφορά την εφαρμογή της ΚΑΠ στα κράτη-μέλη. Και αναφέρθηκε η ευελιξία και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του προγράμματος για τους νέους γεωργούς. Εξού και η ερώτησή μου που προέκυψε από τις πληροφορίες που λάγαμε προηγουμένως. Υπάρχει κατά τη γνώμη σας κάποιος συσχετισμός μεταξύ της εφαρμογής σε επιμερους κρατημέλη ε, περισσότερων ε, μέτρων για τους νέους γεωργούς ε, για την ηλική ε, ανανέωση. Υπάρχει συσχετισμός αυτών των μέτρων με τους δείκτες που μας αναφέρατε. Σίγουρα υπάρχουν μεγάλες διαφορές Υπάρχουν μεγάλε διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών που οφείλονται και σε διαφορετικέ παραδόσει και τρόπου παραγωγή, αλλά υπάρχει σχέση μεταξύ των μέτρων και των δικτών. Γιατί αυτό θα είναι σημαντικό συμπέρασμα που θα ληφθεί υπόψη στη συζήτηση για το μέλλον τη γεωργική πολιτική. Ευχαριστώ. Εγώ έχω μια ερώτηση ω προ την επιλογή των περιφερειών και των χωρών που συμπεριλάβατε στον έλεγχο. Ε, και τι ακριβώς ελέγξατε, τι είδους εκμεταλλεύσεις, ε, μεγαλύτερες, μικρότερες ή χώρες στις οποίες υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη συνέχιση, αν υπάρχει πρόσβαση στο κεφάλαιο, οπότε είναι προσοδοφόρα η συνέχιση της γεωρικής παραγωγής. Γιατί στη Βαρμία Μαζουρία ο μέσος όρος είναι 35 εκτάρια γεωρική εκμετάλλευση. Ενώ ανατολικά της Πολωνίας είναι 4-5 εκτάρια. Οπότε διαφορετικά θα ήταν τα συμπεράσματα, λαμβάνετε υπόψη άλλε περιφέρειες στον έλεγχό σα. Η επιλογή των περιφερειών προδικάζει κατά κάποιο τρόπο τα αποτελέσματα της έκθεσης. Με ποιο κριτήριο επιλέξετε τις συγκεκριμένες περιφέρειες, λοιπόν. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της ε, Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Πάσκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και εσάς κύριε Βοσικόφσκι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να ανταλλάξουμε απόψεις για τη σημαντική αυτή ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου που έχει να κάνει με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους νέους γεωργούς. Εμείς συμφωνούμε σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο ότι η αποτελεσματική υποστήριξη προς τους νέους γεωργούς είναι πάρα πολύ σημαντική αν πρέπει να καταφέρουμε τελικά να υποστηρίξουμε τον γεωργικό τομέα, αυτό θα πρέπει να γίνει σαφώς και μέσω των νέων γεωργών. Η έκθεσή σας ασχολείται με όλα τα διαφορετικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν, ότι θα πρέπει ε, να αυξηθούν τα μέτρα στήριξης των νέων γεωργών, να δημιουργηθεί ένα νέο καθεστώς στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα για την υποστήριξη των νέων γεωργών, στα πλαίσια των άμεσων ενισχύσεων. Ε, καλωσορίζουμε τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου, αρκεί βέβαια να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μην προδικάζουν βέβαια το πολιτικό πλαίσιο το οποίο θα προκύψει μετά το 2020. Παρ' όλα αυτά θα θέλαμε και εμείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποθετηθούμε για κάποια σημαντικά ζητήματα που έθεσε το Ελεκτικό συνέδριο και τα οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να τονίσουμε και για τα οποία θα πρέπει να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Πρώτον, να τονίσω ότι όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή ε, του ελεγχού σα και όσον αφορά την έλλειψη τη στοχοθέτηση, στον πρώτο πυλώνα στι ε, ενισχύσει των νέων γεωργών, μπορεί να προβλέπονται εδώ πέρα νέε πληρωμέ για τους νέους γεωργούς, οι οποίοι όμως πρόσφατα ήδη έχουν εγκατασταθεί ή δημιούργησαν μια οργική εκμετάλλευση. Αυτό ισχύει για μια περίοδο πέντε ετών. Ακριβώ για να αντιμετωπίσουμε τις ειδικέ οικονομικές ανάγκες των νέων αυτών γεωργών, οικονομικές ανάγκες που προκύπτουν μετά τη δημιουργία της οικονομικής εκμετάλλευσης. Ξέρετε ότι αυτή η πρώτη χρονική περίοδος είναι ιδιαίτερη κρίσιμη και χαρακτηρίζεται από υψηλέ οικονομικές ανάγκες. Τονίζω λοιπόν ότι αυτή η ενίσχυση προς τους νέους γεωργούς δεν δίνεται μόνο στα πλαίσια της πληρωμής για των νέων γεωργών, δεν είναι μεμονωμένη ενίσχυση, αλλά είναι μία πληρωμή υπέρχεται ως συμπλήρωση προς τη βασική πληρωμή ή αυτό το οποίο ονομάζουμε green payment, την ε, ενίσχυση η οποία δίνεται για το greening προς τους νέους γεωργούς. Αυτό ισχύει ήδη για την υφιστάμενη περίοδο 2005-2020 και εν γέννη 15 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθούν σάμες ενισχύσεις στους νέους γεωργούς Έξι φορές δηλαδή το ποσό των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ που αναφέρετε εσείς στη δική σας την έκθεση. Όσον αφορά την άπτυξη της υπαίθρου, η ειδική έκθεση του συνεδρίου επικεντρώνεται στα συγκεκριμένα μέσα και εργαλεία που έχουμε για την εγκατάσταση των νέων γεωργών Εν προκειμένου όμω δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα οι νέοι γεωργοί μπορεί να αποφεληθούν από πολλέ άλλε ενισχύσει που καλύπτουν τη μεταφορά γνώσεων, ενημέρωση, πληροφόρηση, διαχείριση των γεωργικών εκμετάλλευσεων και πολλέ άλλε υπηρεσίε. Μπορούν λοιπόν οι νέοι γεωργοί να αποφεληθούν από διάφορα μέτρα του δεύτερου πυλώνα προκειμένου να καταφέρουν με επιτυχία να εγκαταστήσουν αυτή τη νέα γεωργική δραστηριότητα υπολογίζεται ότι 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ δημοσίων δαπανών που έχουν προγραμματιστεί στα πλαίσια της τρέχουσας περίοδου για τον ειδικό αυτό στόχο της διευκόλυνσης των νέων γεωργών στον γεωργικό τομέα πρόκειται να δοθούν. 180.000 νέοι γεωργοί θα υποφεληθούν από το μέτρο αυτό. Το μέτρο αυτό εγκατάστασης δημιουργεί μια οικονομική βιωσιμότητα για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσω πολλών διαφορετικών μέσων ένα μέσο έχει να κάνει με τις ειδικέ συνθήκες που υπάρχουν, δηλαδή η υποστήριξη μπορεί να δοθεί με βάση τις συγκεκριμένε συνθήκες που υπάρχουν για τη γεωρική εκμετάλλευση, μπορεί να δοθεί με βάση τη έγκριση ενό επιχειρηματικού σχεδίου, μπορεί να δοθεί σε έναν ελάχιστο αριθμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Υπάρχει λοιπόν μια στοχοθέτηση όσον αφορά αυτή την υποστήριξη. Πέρα από αυτό, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την υποχρεωτική εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας, τα οποία καθορίζονται από τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της συντρέχουσας αυτής αρμοδιότητας διαχείρισης του δεύτερου πυλώνα. Όσον αφορά το ζήτημα του συντονισμού, νομίζω ότι το ελεκτικό συνέδριο επέκρινε την έλλειψη συντονισμού μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Πρέπει ως προς αυτό να τονίσω ότι κατά την άποψή μας υπάρχει μια εγγενή συμπληρωματικότητα ανάμεσα στις δύο αυτές μορφές υποστήριξης. Και οι δύο αυτές μορφές υποστήριξης βέβαια προσπαθούν να πετύχουν διαφορετικούς στόχους. Στον πρώτο πυλώνα προσπαθούμε να δώσουμε επιπλέον ενισχύσεις για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο που φτάνει έως και την πενταετία και είναι συμπληρωματικές οι ενισχύσεις αυτές σε σχέση με την υποστήριξη που έχουμε στο δεύτερο πυλώνα, μια κατοποκοπήν υποστήριξη βασικά που βοηθά τον νέο γεωργό να στήσει μια νέα γεωργική εκμετάλλευση και κατά αυτόν τον τρόπο να προσχωρήσει στο γεωργικό τομέα. Πέρα από αυτό και πάντα ως προς την πληρωματικότητα θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν στην διάθεσή τους πολλά, με, μέσα για να πετύχουν τον καλύτερο δυνατό συντονισμό μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Τέλος, να σας πενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απόλυτα δεσμευμένη να αυξήσει τις επιδόσεις της και θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλη την αξιολόγηση που γίνεται σε νοσιακό επίπεδο. Να αναφέρω επίσης και να ενημερώσω ουσιαστικά την Επιτροπή Γεωργίας για τις επιπτώσεις της κοινή γεωργικής πολιτικής όσον αφορά την ανανέωση των γενναιών. Θα κάνουμε μια συγκεκριμένη αξιολόγηση η οποία θα ξεκινήσει στα τέλη του 2017 και όπου θα βλέπουμε ακριβώς πώς η κοινή γεωργική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την πραγματική ανανέωση των γενναιών. Θα εξετάσουμε όλα τα μέσα τα οποία έχουμε τόσο στον πρώτο όσο και στο δεύτερο πυλώνα για του νέου γεωργού χωρίς να αφαιρόμαστε όμως μόνο και αποκλειστικά στην υποστήριξη εγκατάστασης. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τη σφαιρική αυτή αξιολόγηση για να δούμε ποια είναι η γενικότερη επίπτωση των μέτρων υποστήριξης στα πλαίσια της κοινή διοργικής πολιτικής όσον αφορά τον απότερο στόχο της ανανέωσης των γενεών. Και μία ακόμη ερώτηση. Ακόμη Η στρεματική ενίσχυση. Ε, επηρεάζουν ε, τη μεταβίβαση γης στους νέους γεωργούς και με ποιο τρόπο. Γιατί φαντάζομαι κάποιος που θέλει να γίνει ιδιοκτήτης τον ενδιαφέρει πρόσβαση σε επιπλέον κεφάλαιο, σε επιπλέον μέσα. Επίση, μπορεί να θέλει ο νέος να παραμείνει στην Γεωργία, αλλά η αραβωνιαστικιά του να μην θέλει, να μπορεί να βρει σύζυγο ως Γεωργός γιατί πραγματικά είναι δύσκολη η γεωργική δραστηριότητα, επηρεάζεται από τι κοινωνικέ συνθήκε και μερικέ φορέ οι δυσκολίε είναι και εξωτερικέ. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα, μια και έχω τη δυνατότητα. Ευχαριστώ θερμά τους ε, ευρωβουλευτές για τη συμμετοχή τους στη συζήτηση, για τις ερωτήσεις που έθεσαν, για τις σκέψεις που παρουσίασαν και χαίρομαι ιδιαίτερος που η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου αποτέλεσε τη βάση για τόσο ενδιαφέρουσα εισαγωγική συζήτηση για το θέμα αυτό. Γιατί όλοι έχουμε επίγνωση ότι το θέμα ξεκινά εδώ, είναι, ήταν το σημείο αφετηρίας αυτή τη συζήτηση ε, και σίγουρα το θέμα θα μας απασχολήσει και στο μέλλον ε, για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ε, καταρχήν κάτι που προκύπτει από τα έμεσα συμπεράσματα του ελέγχου. Το πρόβλημα των νέων γεωργών, όπως ανέφεραν και πολλοί ευρωβουλευτές, θα πρέπει να το δούμε ε, από τη σκοπιά του συνόλου της κοινή γεωργικής πολιτικής. Τι γίνεται, δεν έχετε διερμηνία. ο English. Ε. I can repeat in English my... Μπορώ να τα επαναλάβω και στα αγγλικά. Continue Polish. Yes. The, I'd like to, to... Uh- Επαναλαμβάνω το κεντρικό συμπέρασμα ότι το πρόβλημα των νέων γεωργών θα πρέπει να το εξετάσουμε υπό γενικότερη σκοπιά, γιατί αφορά το σύνολο της κοινή γεωργική πολιτικής και αφορά ολόκληρο το μέλλον της κοινή γεωργική πολιτικής το θέμα των νέων γεωργών. Και η συζήτηση για τη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική, το δεν αρκεί να την περιορίσουμε στην επόμενη επταετία. Θα πρέπει να έχουμε ένα όραμα για το τι μορφή θέλουμε να έχει η Ευρωπαϊκή Γεωργία μετά από 30 χρόνια. Τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Γεωργία το 2050. Δεν θα πρέπει στη συζήτηση για το μέλλον τη κοινή γεωργική πολιτικής να περιοριστούμε χρονικά στον πολύ χρονικό ορίζοντα. Ε, ως ε, μέλος του ελεκτικού συνεδρίου ε, δεν μπορώ να δώσω απάντηση για το αν η μείωση του αριθμού των ε, αγροτών θα πρέπει να μας χαροποιεί να μας θλίβει. Γιατί υπάρχουν και στη γεωργία τεχνολογικές εξελίξεις, υπάρχουν μικρές ή μεγάλες καλλιέργειες. Θα πρέπει όμως να δώσουμε την απάντηση στο πώς φανταζόμαστε εμείς την Ευρωπαϊκή Γεωργία το 2050. Τι μόρφη θα πρέπει να έχει. Και αυτή η μείωση στα 10 εκατομμύρια θα πρέπει να αναχαιτιστεί ε, όταν πριν από 20 χρόνια άρχισα να ασχολούμαι με την πολιτική και μου έθεταν το ερώτημα, θα έλεγα ναι, πρέπει να αναχαιτήσουμε την ε, φθήνουσα αυτή πορεία του αγροτικού πληθυσμού. Ε, κατά τη γνώμη μου, η έλλειψη οράματος στη γεωργία και από το παρελθόν είναι αιτία ε, πολλών αποτυχιών ευρωπαϊκών πολιτικών και όχι μόνο κάποιων ελλείψεων και αποτυχιών της κοινή ζωρικής πολιτικής. Θα πρέπει να έχουμε πολύ πιο μακροπρόθεσμο όραμα σε όλες μας τις πολιτικές. Επίσης, ε, ε, Σίγουρα δεν θα πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η στήριξη είναι περιττή επειδή δεν είναι αρκετά αποτελεσματική και θα πρέπει να την καταργήσουμε. Το αντίθετο, η κατάσταση στην Ήπεθρο είναι τραγική. Γι' αυτό και χρειάζεται καλύτερη ενίσχυση και καλύτερα στοχοθετημένη ε, και προσανατολισμένη ενίσχυση. Σε καμία περίπτωση δεν είναι περιττή αυτή η ενίσχυση στους νέους γεωργούς. Η κυρία Εράς και η κυρία Αγγιλέρα ε, μίλησα για κάποιες επικρίσεις προς ε, συγκεκριμένες χώρες ή συγκεκριμένες περιφέρειες, όπως τα Ανταλουσία. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλάβετε την έκθεσή ως ένα ανθολόγιο επικρίσεων ε, κατά κρατών, περιφερειών ή συγκεκριμένων γεωργών. Όχι. Το πρόβλημα δεν είναι σε επίπεδο γεωργών. Το πρόβλημα είναι στο επίπεδο της συλλογική της παρέμβασης. Και εγώ όσο ήμουν Ευρωβουλευτής ε, συμμετείχα στη συζήτηση τι μορφή θα πρέπει να έχει το καθεστώς ενισχύσεων ε, με βάση τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ένα επίπεδο θετικών αποτελεσμάτων και δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στην ερώτηση αυτή γιατί δεν έχουμε δείκτες, δεν έχουμε τρόπους μέτρησης για να δούμε σε, σε τι βαθμό η συνδρομή αυτή, η ενίσχυση συνέβαλε στη βελτίωση της ε, ηλικιακής δομής. Από τα γενικά στοιχεία μάλλον δεν συνέβαλε αυτή η σύνδρομη. Αλλά μπορεί αν δεν είχαμε αυτή την ενίσχυση να ήταν πολύ χειρότερη η ηλικιακή ανανέωση, πολύ χαμηλότερο το ποσοστό. Ο κύριος Κούσμιουκ μίλησε για μετρήσιμους δείκτες. Φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα κριτήρια SMART, δηλαδή θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα, μετρήσιμα, εφικτά, ρεαλιστικά και χρονικά προσδιορισμένα. Δέκα δισεκατομμύρια ε, ευρώ έχουν δαπανηθεί για τη στήριξη των νέων γεωργών. Αλλά δεν έχουμε συγκεκριμένους δείκτες, μετρήσιμους, εφικτούς, ε, δυστυχώς δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα χωρίς να έχουμε τέτοιους συγκρίσιμους δείκτες. Επίσης υπήρχε πρόβλημα με τη λογική της παρέμβασης. Αυτή θα πρέπει να τη διορθώσουμε στο μέλλον. Από την Πολωνία δόθηκε το παράδειγμα στην έκθεση ότι λαμβάνει ενίσχυση ε, που έχει πάνω από 513 εκτάρια. Ναι, ωραία που έλαβε την ενίσχυση. Δεν έχω πρόβλημα να λαμβάνει ενίσχυση και ένας γεωργός με πολλά στρέμματα. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει το κράτος που έδωσε ενίσχυση και σε τέτοιο γεωκτήμονα Γιώργο. Θα πρέπει όμως να δούμε τη λογική της ενίσχυσης και σε τι βαθμό η ενίσχυση συμβάλλει στη βελτίωση της ε, ηλικιακής ανανέωσης. Φαίνεται ότι σε κανένα βαθμό δεν επηρέασε η βοήθεια ούτε στην ανάληψη της ε, γεωργικής εκμετάλλευσης από τον νέο Γεωργό, ούτε στην απόφαση το κατά πόσο θα παραμείνει στην εκμετάλλευση. Άλλοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την απόφαση, αυτή τη μεταβίβαση και όχι η συγκεκριμένη στήριξη. Οπότε θα πρέπει η λογική της παρέμβασης πραγματικά να συμβάλλει στη βελτίωση της δομής, της ηλικιακής δομής των γεωργών. Πολύ εύστοχα επισημάνατε ε, το συσχετισμό του συστήματος ε, ασφάλειας. Δεν σημείωσα με λεπτομέρειες τα ονόματα. Νομίζω ο κύριος Ντες το ανέφερε και ίσως και κάποιοι άλλοι ευρωβουλευτές. Ε, τώρα σίγουρα το, θα πρέπει να το συνδέσουμε με το σύστημα ε, ε, ασφαλιών για το ότι έχουμε τόσους πολλούς ε, ηλικιωμένους γεωργούς. Και σίγουρα η βοήθεια στους νέους γεωργούς, όλους παραδόξως, ισοδυναμεί έμεσα με βοήθεια και σε ηλικιωμένους γεωργούς. Είναι περίπλοκο βέβαια αυτό το θέμα και θα χρειαστούν και πολλές δραστηριότητες για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ο κύριος Καλινόφσκι μίλησε για την ευελιξία και εδώ πραγματικά διαπιστώνουμε ένα πρόβλημα είναι καλό να εφαρμόζουμε το ίδιο φάρμακο σε διαφορετικές ασθένειες, γιατί η κατάσταση μεταξύ των κρατών μελών είναι πολύ διαφορετική. Αν στη Γερμανία, για παράδειγμα, έχουμε τους 6,5% μόνο τους ηλικιωμένους γεωργούς, ενώ στην Πορτογαλία είναι 50% των γεωργών ηλικιωμένοι, δεν μπορούμε τα ίδια μέσα και τους ίδιους μηχανισμούς να τους εφαρμόζουμε σε δύο χώρες που έχουν τόσο διαφορετικές καταστάσεις χρειάζεται μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών και θα πρέπει να τη βρούμε αυτή τη διαφοροποιημένη προσέγγιση. Επίσης, ε, πρόσβαση στην αγορά γη. Αυτό το πρόβλημα το εντοπίσαμε και με την έκθεσή μας. Το είπαν ο κύριο Ροπέ, ο κύριος Χόισλινγκ, ότι δύσκολα έχουν πρόσβαση στην αγορά γη. Και ίσω, ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι είναι το πρόβλημα της γης. 60% των νέων γεωργών από την έρευνα που κάναμε ε, μας είπαν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για αυτούς είναι η γη. Έχουν και πρόβλημα με την πρόσβαση στο δανεισμό, στο κεφάλαιο, αλλά για, τους νέους γεωργούς η πρόσβαση στη γη είναι το πιο δύσκολο πρόβλημα και στην Πολωνία εγκρίθηκε ένας νόμος πολύ επίμαχος που ε, περιόρισε την πρόσβαση στη γη σε άτομα που δεν ασκούν γεωργικές δραστηριότητες. Ε, ίσως θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση ώστε να μπορεί ο Γεωργός να έχει πρόσβαση στην αγορά της γης. Γιατί οι νέοι Γεωργοί χρειάζονται εκτάσεις γεωργικές για να αναπτύξουν τις γεωρικές δραστηριότητες. Και θα πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους να τους διευκολύνουμε για να μπορέσουν να αγοράσουν γεωρικές εκτάσεις. Φαίνεται ότι υπάρχει επίγνωση του προβλήματος ε, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είχαμε συνεργασία και κατά την εκπόνηση έκθεση. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να μεταρρυθμιστεί αυτό το σύστημα στήριξης των γεωργών. Η στήριξη όμως είναι απαραίτητη γιατί διαπιστώνουμε ότι ε, οι νέοι γεωργοί είναι το 20% του γεωργικού πληθυσμού, σε αντίθεση με τους νέους γενικά που είναι 50% του εργατικού δυναμικού σε άλλους κλάδους. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να βελτιώσουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση και την παρουσία των νέων γεωργών στη Γεωργία. Ευχαριστώ κυρία Χόιμπουχ. Πολύ σύντομα μας παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχά, μπορούμε να βάλουμε τα δύο μικρόφωνα από το τραπέζι πάνω σε εσά, το Προεδρείο. Ακούσαμε προηγουμένω ότι με του νέου γεωργού δεν θέλουν να πάνε οι γυναίκε να ζήσουν μαζί του, ότι έχουν ένα πρόβλημα εδώ. Όμω, οι νέοι γεωργοί έχουμε πει και εμεί ότι είναι και καινοτόμοι, αλλά και ότι ο αριθμός νέων γυναικών είναι υψηλότερος. Οπότε να μην βάζουμε τις γυναίκες εδώ πέρα να τις κατηγορούμε. Αυτό θέλω να τονίσω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, ε, πρέπει να απαντήσω πρώτα στον ε, πρόεδρο που ρώτησε αν οι ενισχύσεις περιόρισαν ε, την μεταβίβαση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των αγροκτημάτων. Δεν έχουμε στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ή να διαψεύδουν αυτή τη διαπίστωση. Επίσης, επίσης, δεν μπορούμε να απαντήσουμε ποια είναι καλύτερη ενίσχυση του πρώτου ή του δεύτερου πυλώνα. Σίγουρα έδωσαν κάποια ναύσματα τέτοιες ενισχύσεις, αλλά ε, μόνο 7% των γεωργών επωφελήθηκε από τις ενισχύσεις όταν υπήρχαν μόνο στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα. Πολύ μικρός αριθμός λοιπόν. Και ο πρώτος πυλώνας ε, είναι πολύ πιο δίκαιος για τους περισσότερους γεωργούς, αλλά δεν μπορούμε να τον συνδέσουμε με κάποια αποτελέσματα στην γεωργική διαχείριση. Θα πρέπει στο μέλλον να δούμε πώς θα οργανώσουμε καλύτερα την κατάσταση. Σας ευχαριστώ θερμά γιατί πραγματικά δημιουργήσατε ιστορία, προηγούμενο, γιατί πρώτη φορά ε, υποβάλλεται ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Υπάρχει η συνήθιση ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, αλλά κατά τη γνώμη μα είναι σημαντικό να, υποβάλλω, να παρουσιάζονται και οι ειδικέ εκθέσει του Ελεγκτικού Συνεδρίου στι ε, συγκεκριμένε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Κάτι τέτοιο έγινε και στην Αλλιευτική Επιτροπή, στην Επιτροπή Αλίας, όπου παρουσιάσαμε την ειδική έκθεση για την Αλία. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να παρουσιάζονται αυτές οι ειδικέ εκθέσεις στις κοινοβουλευτικέ επιτροπές που ασχολούνται με το θέμα που είναι το αντικείμενό του. Σας ευχαριστώ θερμά γιατί πραγματικά συμβάλλετε στην μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής και σας ευχαριστώ θερμά για τη θερμή υποδοχή που επιφυλάξατε στην έκθεση. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ήταν πολύ καλή απόφαση να έρθετε στην Επιτροπή μας για να μας παρουσιάσετε την ειδική έκθεση και χαίρομαι για την αλλαγή αυτή στην πολιτική του ελεκτικού συνεδρίου γιατί όλοι θα βγούμε κερδισμένοι από μια τέτοια ανταλλαγή απόψεων. Γενικώ πάντως οι νέοι γεωργοί βλέπουν θετικά την στήριξη. Τώρα για τους μηχανισμούς και τη μορφή που θα λαμβάνει ίσως και τον τρόπο εφαρμογής στο μέλλον ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε και στη συνέχεια πιο διεξοδικά. Σας ευχαριστούμε και πάλι θερμά και επειδή έχουμε καθυστερήσει να περάσουμε αμέσως στο επόμενο σημείο και να δώσω το λόγο στην κυρία Ντελαέ. Ευχαριστούμε και πάλι θερμά κύριε Βοητσεχόφσκη. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Ντελαέ, που θα μας παρουσιάσει τη γνωμοδότησή της για τον ορισμό, παρουσίαση, επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση ονομάτων ε, ενοπνευματοδών ποτών στην παρουσίαση και την ε, ετικετοθεσία ε, άλλων τροφίμων και την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών. Δεν θα κάνω εγώ άλλη παρουσίαση, είστε αρμόδιοι κυρία Ντελέ και θα μας την κάνετε πολύ καλύτερα από μένα αυτή την ενημέρωση. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το κείμενο που σας παρουσιάζω σήμερα είναι μια γνωμοδότηση για ένα σχέδιο έκθεσης της κυρίας Πιλάρα Γιούζο από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Μήπως να αφήσω πρώτα τους συναδέλφους να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, Πρόκειται για την πρόταση κανονισμού για τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμαση των αλκοόλικων πολιτών. Δεν διαβάζουν υπόλοιπο τίτλων ιδιαίτερα μακροσκελή. Τα συστήματα προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων αποτελούν ε, πολύ σημαντική πρόκληση και σημαντικό διακύβευμα και για την δική μα την ενωσιακή εμπορική πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί όχι μόνο να καταφέρει να προστατεύσει τα σήματα ποιότητα στην εξωτερική αγορά, αλλά και να δώσει κίνητρα στις τρίτες χώρες να αρχίσουν και αυτά να χρησιμοποιούν στις δικές τους χώρες, στη δική τους επικράτεια, αντίστοιχα σήματα ποιότητα. Όσον αφορά τον τομέα των αλκοόλουχων ποτών, ξέρετε ότι είναι ένα τομέα κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των πολύ μεγάλων εξαγωγών περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ, σε 10 δισεκατομμύρια ευρώ αντιστοιχείο το των εξαγωγών για τα αλκοολούχα ποτά και απασχολούνται περίπου 1 εκατομμύρια άνθρωποι στον τομέα αυτό. Πρόκειται λοιπόν για έναν πολύ σημαντικό κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, να υπενθυμίσω ότι πέρα από ένα απλό προϊόν κατανάλωσης, τα αλκοολούχα ποτά αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη τεχνογνωσία, σε συγκεκριμένους πολιτισμούς, νοοτροπίες, σε έναν ευρωπαϊκό πολιτισμό ο οποίος εξάγεται προς τα έξω. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε εμείς να επεξεργαστούμε τις τροποποιήσεις που μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά τον τελευταίο κανονισμό, τον 110 του 2008, ο οποίος έπρεπε και αυτός να δραμονιστεί μετά τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Στην πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξυγχρονίζει τον κανονισμό αυτό και είμαστε υπέρ του εξυγχρονισμού αυτού, αλλά έρχεται και δημιουργεί νέα προνόμια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων. Κάνει επίση ουσιαστικέ αλλαγέ στον κανονισμό αυτό και οι τροποποιήσει αυτέ μα προβληματίζουν. Εφτά αλλαγέ έχω εντοπίσει. Θα σα δώσω δύο πιο συγκεκριμένα παραδείγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταργεί το παράρτημα 3, όπου έχουμε τι γεωγραφικέ ενδείξει και αντικαθιστά το παράρτημα αυτό με ένα μητρό. Επί της αρχής δεν θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει πάρα πολύ ασαφής με αυτό το μητρό. Και παράλληλα έχει, δίνει στον εαυτό της την αρμοδιότητα να αλλάζει μέσω εκτελεστικών πράξεων αυτό το μητρό, να επιφέρει αλλαγές. Πρώτο πρόβλημα λοιπόν που εντοπίζουμε σε αυτό το σημείο. Δεύτερον, όσον αφορά την απαγόρευση μετάφρασης των γεωγραφικών ενδείξεων σε διαφορετικές διαφορετικά συστήματα γραφής, όπως γράφουμε από αυτά που έχουμε σε σχετικές χώρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει τη μετάφραση των γραφικών ενδείξεων μόνο μέσω κατεξοδότηση πράξεων, ενώ στο προηγούμενο κείμενο είχαμε την δυνατότητα αυτόματης και συστηματικής μετάφρασης των γραφικών αυτών ενδείξεων. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική πίσω από τις αποφάσεις αυτές. Δεν νομίζω ότι επιτυχάνεται κάποια απλούστευση, αν αυτό τελικά θέλει να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω αυτών των τροποποιήσεων. Η απλούστευση ενός κειμένου πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, όταν το ίδιο το κείμενο αυτό εφαρμόζεται και έχει γίνει αποδεκτό από διάφορους κλάδους. Η πρόταση επίσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να περιοριστεί στον εξεχρονισμό του κειμένου του 2008, θα πρέπει να περιορίσει όσο τον το περισσότερο οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση και δεν θα πρέπει να δημιουργεί νέες αρμοδιότητες, ιδίως όταν αυτές επηρεάζουν τις γεωγραφικές ενδείξεις. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο υπέβαλα αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και θα πρέπει να σας πω ότι το ζήτημα αυτό είναι ένα ζήτημα κυρίως τεχνικό. Δεν είναι λοιπόν λογικό η Επιτροπή, η δικιά μας Επιτροπή Γεωργίας, να είναι απλώς μια γνωμοδοτική επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό να υποθεί αυτό. Να επιθυμίσω επίση στου αδέλφου ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή για έναν τεχνικό κανονισμό που έχει να κάνει με την επισήμανση. Δεν πρόκειται για έναν κανονισμό που θα έχει να κάνει με την υγεία και την προστασία των καταναλωτών από τους κινδύνους που συνδέονται με την υπερβολική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Σας ζητώ λοιπόν μέσω των τροπολογιών σας να επικεντρωθείτε κι εσείς περισσότερο στο κείμενο του 2008. Θα είμαι στη διάθεσή σας και εγώ και οι συνεργάτες μου για οποιοδήποτε ζήτημα θέλετε να θίξετε στα πλαίσια της γνωμοδότησης αυτής. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η Παρασκευή 14 Ιουλίου η επόμενη Παρασκευή δηλαδή, η ερχόμενη Παρασκευή. Ελπίζω ότι ήμουν να σαφή στην τοποθέτησή μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ταραμπέλα που είναι και σκιώδης ηγετής. Ευχαριστώ Πρόεδρε η κυρία Δελαέ. Υπενθύμησε αρχικά τη σημασία του κλάδου αυτού για την Ευρώπη. 8% δηλαδή του συνόλου των εξαγωγών αυτού του κλάδου της Ευρώπης, δηλαδή των ακολούχων για τον κανονισμό 110-2008 ικανοποιούσε σε μεγάλο βαθμό τους ε, φορείς του κλάδου και να πω επίσης ότι το 4 2 αυτής της ε, προσυμφωνίας αποτέλεσε την ε, νομική βάση η οποία βοήθησε αυτή την νομοθεσία ώστε να βρει μια λύση όσον αφορά την ποιότητα και τα ποσοτικά στοιχεία ώστε η παραγωγή αυτών των αλκοολούχων ποτών να γίνεται με προϊόντα γεωργικής προέλευσης. Η κυρία Τελαέ, ελπίζω να μην αλλάξει περιβολικά το κείμενο, γιατί νομίζω ότι πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση, απλά και μόνο θα αναφερθώ σύντομα σε κάποια στοιχεία σημαντικά που μου φαίνονται και είναι τρία καταρχάς να στηρίξουμε τις τεχνικές διορθώσεις όσον αφορά το άρθρο 2 που αναφέρεται στον 110.008 όπως επίσης και τη δυνατότητα του άρθρου 8 να μεταφράζονται οι σημάτσεις. Νομίζω ότι για τις ε, κατεξοδότητες πράξεις νομίζω ότι αυτό είναι θέμα λογικής. Μετά για το άρθρο 12 σε σχέση με τον κανόνα πρόελευση. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να ε, οδηγήσει σε σφάλμα τον καταναλωτή, γιατί η προέλευση δεν καθορίζεται πάντως σύμφωνα με τον τελευταίο τόπο μεταποίηση του προϊόντο, Αν πάνω από το 85% του προϊόντο ε, αποτελείται από αλκοόλ από την ίδια χώρα ή από την ίδια περιοχή. Τι θα πούμε, α πούμε, οι Σκοτσέζοι αν έχουμε βελγικό ουίσκι με 80% σκοτσέζικο ουίσκι, αλλά προστίθεται κάποια αρωματικά εδώ στι Βρυξέλλε. Δεν είναι σκοτσέζικο ουίσκι, ξεκάθαρα. Οπότε υπάρχουν επιφυλάξει. Επίση, έχουμε βολή σε σχέση με τα μείγματα που προτείνονται και νομίζω ότι αυτά προτείνονται είναι λιγότερο σαφή από αυτά που προτείνει η Κομισιόν. Οπότε θα πρέπει να το συζητήσουμε και θα πρέπει να βρούμε μια λύση. Τρίτο σημείο, νομίζω ότι είναι σημαντικό να αντικαταστήσουμε τον όρο προστασία με τον καταγραφή. Γιατί ο όρος προστασία όπως προτείνει η Κομισιόν είναι διφορούμενος γιατί υπάρχουν προστατευόμενες γραφικές ενδείξεις που υπόκειται σε διαφορετικούς κανόνες από ότι η γεωγραφική ένδειξη. Και τέλος να πω ότι χαίρομαι που συνεργάστηκα με την συγκέντρια και τους κοιόδε, ώστε να έχουμε τελικά ένα φιλόδοξο και ισόρροπο κείμενο και το οποίο θα διασκεδάζει ανησυχίες και μέσα στο πολύ. Ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα τους κέντες ε, να μιλήσουν για δύο λεπτό καθένας και οι υπόλοιποι για ένα λεπτό καθένας. Παρακαλώ κύριε Φλάνναγκαν. Ε, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ελπίζω να το αφήσουμε για αύριο γιατί αύριο θα συναντήσουμε μικροσώπους, Microsoft του κλάδου. Όμως να τονίσω ότι κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η ρύθμιση είναι πιο λογική από το χάος. Και εγώ ε, ξέρω τι γίνεται με την κάναβη και με τα ουίσκι σχετικά. Δεν ξέρω λοιπόν ε, κατά πόσο τέλο πάντων ε, τον υπάρχει ένα στην καλλιέργεια, να είναι γιατί αν δεν θα ήταν καλή ιδέα, ίσω να μην χρειαζόταν να το κάνουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη από ό,τι είπαν οι συναδέλφοι, ανακύπτει ότι ο κλάδο αυτό είναι σημαντικό και έχει επιπτώσει στην οικονομία, στι θέσει εργασία, στις εξαγωγές, 8% των αστυνομικών υλικών εξαγωγών, όπω είπαμε. Οπότε ο 110-2008 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο κίνηση και να προσαρμοστεί χωρίς μεγάλε τροποποιήσει. Όμως, να κάνω μια σκέψη για το τι σημαίνει το να εφαρμόσουμε στη συνέχεια και πώ εφαρμόσουμε στη συνέχεια του κανονισμούς. Γιατί αν δεν υπάρξει συντονισμό σε διάφορα θεσμικά επίπεδα, κοινοτικό, εθνικό, τοπικό, θα μπορούσαν να υπάρξουν δυσάρεστε καταστάσει, ιδιαίτερα όταν έχουμε ομονιμία μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών. Ας πούμε, να επενθυμίσω το τι συνέβη στη δική μου την ε, περιοχή της Βενετίας με το κρασί. Σε μια περιοχή το, το ΚΑΙ αφαιρέθηκε επειδή ακριβώς είχε την ατυχία να είναι ομώνυμο, να έχει το ίδιο όνομα, με ένα άλλο προϊόν, το οποίο προστατεύεται, είναι προστατευμένο στην Ουγγαρία. Οπότε θα πρέπει να προσέχουμε λοιπόν την εφαρμογή των κανόνων ώστε η θεραπεία να μην είναι χειρότερη από το κακό. Θα πρέπει να δούμε επίσης και τις ανάγκες των παραγωγών και την ανάγκη προστασίας των καταναλωτών. Και αναφέρομαι εδώ ιδιαίτερα στην διατήρηση ενός υψηλότατου επίπεδου ποιότητας παραπέμποντα, α πούμε, στο άρθρο 3, που αναφέρει ότι το αλκοόλ το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασχολή παρασκευή αυτών των προϊόντων θα πρέπει να έχει γεωρική προέλευση. Αυτό νομίζω είναι βασικό. Όπως επίσης για τι πληροφορίε θα έλεγα ότι είναι βασικό να αναφέρονται στη σήμανση οι προελεύσεις των κυριοτέρων στοιχείων που απαρτίζουν αυτό το προϊόν. Ευχαριστώ. Κυρία Εράνς, ευχαριστώ. Για την κυρία Τελε και για μένα το θέμα είναι πολύ σημαντικό και για τις χώρες μας το ίδιο ο κανονισμός για τα αλκοόλουχα ποτά. Εγώ θα μιλήσω για τη λίκανση, ε, με το στρογγύλεμα της γεύσης. Είπατε ότι θα, ανάλογα με κατηγορία θα έχουμε τα ανώτατα όρια. Στο παράρτημα 2 όμως λέτε ότι όλα τα προϊόντα θα έχουν ανώτατο όριο 2 γραμμάρια ανά λίτρο. Οπότε έχουμε πρόβλημα. Δεν αφήνουμε ελεύθερο το ανώτατο όριο κάθε κατηγορίας. Θα καταθέσω σχετική τροπολογία και ελπίζω να τη λάβετε υπόψη. Κάθε προϊόν έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, οπότε κάθε προϊόν υπόκειται στην εθνική νομοθεσία και θα πρέπει να σεβαστούμε αυτές τις διαφορετικές εθνικές διατάξεις. Ε, κάνετε κονιάκ ε, στη χώρα σας, μπράντι ή χερές στη δική μου πατρίδα ή τέλο πάντων και άλλα αλκοόλουχα ποτά. Οπότε και οι εθνικέ διατάξει θα πρέπει να γίνουν σεβαστέ, γιατί τα περισσότερα προϊόντα έχουν προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Γι' αυτό και θα πρέπει το γενικό το θέμα της γλύκας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις ε, εθνικές διατάξεις και τους κανόνες που ισχύουν για τις γεωγραφικές ενδείξεις. Αυτά και προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία. Η κυρία Μίλλορ παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα αλκοολούχα ποτά της Ευρώπης έχουν πολύ καλή φήμη, απόλυτα δικαιολογημένα. Ξέρετε ότι στην ε, Γερμανία έχουμε κάποιες πολύ μικρές ε, εκμεταλλεύσεις απόσταξης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να επικεντρωθούμε κυρίως σε αυτές τις μικρές εκμεταλλεύσεις και στις παραδοσιακές ε, μορφές παραγωγής. Χρειαζόμαστε όμως και ένα σύστημα ευρυθμό το οποίο θα προστατεύει τις γεωγραφικές ενδείξεις και κατά την άποψή μας, τουλάχιστον για τη Γερμανία, το προτινόμενο αυτό σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε δύο στάδια είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Και είμαστε διστακτικοί επίσης και για το παράρτημα 3, αυτό το οποίο προτείνεται να γίνει μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι γίνεται και με τη γλύκανση και με την περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Θα πρέπει τα αποστακτήρια, τα οποία δεν προσθέτουν ζάχαρη να μπορούν να έχουν και ανάλογη ετικέτα πάνω στα προϊόντα τα οποία παράγουν. Να υπάρχει πληροφορία αυτή στα πλαίσια, τη πλαίσια επισήμανσης. Σχετική τροπολογία θα πρόκειται να καταθέσουμε για όλα αυτά. Ο κύριος Δαντά. Ευχαριστώ. Το κείμενο είναι πολύ σημαντικό και διαπιστώνουμε πως ε, μέσω κάποιων α, ε, ε, παρεκκλήσεων ή έκτροπο που γινόνται, ε, τα αλκοολούχα ποτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στο επίκεντρο ε, επιθέσεων και κριτικών. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διευκρίνηση των κειμένων και ασφάλεια δικαίου. Αυτό είναι σημαντικό για τις, ε, τις δικαστικές μάχες που θα δώσουμε ε, σε διάφορα μέρη του κόσμου. Θα πρέπει να προστατεύσουμε το σύστημα γεωργικών ενδείξεων που έχουμε εκπονήσει στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Άγνιο. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω εμβαθύνει πάρα πολύ στο κείμενο, αλλά μόνο και μόνο ο τίτλος, η συζήτηση που γίνεται και αυτό που ο κύριο Ταραμπέλα έκανε ένα καμπανάκι να αρχίσει να χτυπάει στο κεφάλι μου. Χρησιμοποίησα τον όρο σκότς, ουίσκι. Υπάρχει μια περιοχή στην Βόρεια Βρετανία που ονομάζεται Σκοτία και Θεωρούν βέβαια ότι το ουίσκι αυτό προέρχεται από την Σκοτία. Δεν τους αρέσει όμως ο όρος σκότς. Θα, περιούσαν, θα προτιμούσαν τον όρο Scottish ουίσκι. Έχουμε επίσης και τον όρο Highland Whisky, Highland Malt. Διαβεβαιώ λοιπόν την εισηγήτρια ότι ε, όλες αυτές οι διαφορετικές παραλλαγές αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που ουσιαστικά σε καμία περίπτωση αυτοί που ζουν βόρεια από τα δικά μου τα σύνορα δεν πρόκειται να παραπλανηθούν από αυτά τα οποία προτείνουμε στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Αντρία. Καταρχήν, ζητώ συγγνώμη από την κυρία Ντελαέ γιατί αποσίαζα κατά την παρουσίαση της γνωμοδότησής. Πάντως τη συγχαίρω για το πόνημά της, γιατί πιστεύω ότι η επικαιροποίηση και ο εξυγχρονισμός του κανονισμού για το αλκοόλουχα ποτά ε, είναι απαραίτητες για να μας επιτρέψουν να προστατεύσουμε καλύτερα τι γεωγραφικές μας ενδείξεις όταν ε, πρέπει να ανταγωνιστούμε άλλα προϊόντα εξοκοινωτικά. Καταρχήν, ένα γενικό σχόλιο. Αυτή τη στιγμή ο κανονισμός κάνει διάκριση μεταξύ των ε, αλκοολούχων ποτών και των συγκεκριμένων αποσταγμάτων. Ε, θα πρέπει να αποφύγουμε αθέμητο ανταγωνισμό, κάτι που μερικές φορές συμβαίνει για το ρούμι. Θα πρέπει να διορθώσουμε τη στρέβλωση του ανταγωνισμού που παρατηρούμε και να προβλέψουμε μέγιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη για τα αποστάγματα. Επίσης, ε, για τις ονομασίες Κύρς και Γκινιόλ θα πρέπει να ε, προστατεύσουμε τις γεωρικές ενδείξεις αυτών των παλιών προϊόντων. Επίσης, για το Σίδρα και το Πουαρέ θα πρέπει να παραταθεί η παρέκκληση ό,τι αφορά την αρωματοποίηση για τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και τέλος ό,τι αφορά την ονομασία κονιάκ όπως αναφέρθηκε. Υπάρχει κίνδυνος ε, να θυγεί ε, η υπόλοιψη αυτού του προϊόντος λόγω ανεξέλεγκτης ε, μεθόδου παραγωγής. Ενώ οι, οι κανόνες ΚΟΑ δεν ισχύουν για τα, για τα αμπέλια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κονιάκ, παρόλο που είναι γνωστή και παραδοσιακή αυτή η μέθοδος παραγωγής. Ευχαριστώ. Είναι με ενδιαφέρον το θέμα, αλλά αυτό θα σας δίνει δικαίωμα να μακρηγορείτε. Ο κύριος αλβέρτες. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ θερμά την κυρία Ντελά για την έκθεσή της. Πολύ σημαντικό το θέμα αναφέρθηκαν διάφορα ζητήματα, όπως το άρθρο 5 για τις κατεξοδότηση πράξης. Θα πρέπει να απορρίψουμε την εκχώρηση τέτοιων αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ορισμός των αλκοολούχων τον κατηγορίες του παραρτήματος 2, σημαντικότημα του κανονισμού που δεν θα πρέπει να αλλάζει με κατεξουσιοδότηση πράξης. Το ίδιο ισχύει και με την προσθήκη νέων κατηγοριών. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Αγγιλέρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ για την εισήγηση του συγγητή. Τη συγγήτρια και λέει η συγγήτρια ότι έχουμε να κάνουμε με έναν κανονισμό τεχνικό για την σήμαση και όχι με έναν κανονισμό για την υγεία και την προστασία των καταναλωτών. Αυτό είναι βασικό να το διευκρινίζουμε γιατί καμιά φορά τα μπερδεύουμε. Κυρία Ντελάγε, να διευκρινίσω κάποια πράγματα και να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Μέσω τροπολογιών επιτρέπεται αναπερίπτωση να μιλάμε για την ζάχαρη. 14 συγκεκριμένε τροπολογίες από αυτού. Με ανησυχεί ιδιαίτερα η 34 για το Χερέθ επειδή η Γλύκας ακριβώς το αφήνει απ' έξω με την τροπολογία αυτή που έχετε καταθέσει για αυτό το προϊόν, για αυτό το μπράντι, το χαρέθ που είναι τόσο σημαντικό για τη χώρα μου. 14 λοιπόν ε, τροπολογίες που οριζούν σε 20 γραμμάρια ένα λίτρο. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν για ποιο λόγο. Δεν πάμε πέραν από ό,τι είχαμε πει στην αρχή, επειδή είχαμε πει ακριβώ ότι το κάθε προϊόν συνοδεύεται από δικέ του πρακτικέ. Γι' αυτό ακριβώ έκαναμε του περιορισμού. Οπότε ελπίζω μέσω των τροπολογιών να μπορέσουμε να λύσουμε κάποια από αυτά τα προβλήματα. Και ξαναλέω, με ενισχύει αυτό ιδιαίτερα, γιατί μπορούμε να αφήσουμε εκτός κάποια πράγματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ ταχύτατος. Να ευχαριστήσω καταρχάς τη συνάδελφο Ντελαέ για την έκθεσή της, η οποία είναι σημαντική γιατί το καθεστώς ε, σήμανση γεωγραφικών ενδείξεων αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης. Έχουμε το 110 2008 σημείο αναφοράς. Η Κομισιόν προτείνει μια συνολική αναθεώρηση και εξυγχρονισμό αυτού του κανονισμού και μέσω κατεξουσιοδότησης ε, ε, πράξεων επιφέρει κάποιες αλλαγές σημαντικές, αλλά νομίζω ότι η πρόταση τη Κομισιόν θα πρέπει να περιορίζεται στον εξοχρονισμό του, κειμένου του 2008 και με τη θέσπιση νέων διατάξεων που θα ενισχύουν ακριβώς τις γεωγραφικές ενδείξει και θα ενισχύουν το τρέχον κείμενο. Και από αυτό θα καταθέσω τροπολογίες, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζει η Κομισιόν την συζήτηση στην Άγκρη μετά από την υιοθέτηση της πρώτης Κομισιόν του Δεκεμβρίου 2016. Ιδιαίτερα επειδή είναι η πρώτη φορά όπου υπάρχει μια ε, γεωργική νομική βάση όσον αφορά τα αλκοολούχα, τα οποία έχουν σημαντική προσταμινή αξία στον γεωργικό τομέα και αποτελούν και το στρατηγικό στον τομέα αυτό. Ο οργανισμό 110 ήταν αποτελεσματικό και παρήχε αρκετή ανάπτυξη και θέση εργασία στον κλάδο. Πρέπει όμω να ευθυγραμμιστεί και αυτό ακριβώ προτείνουμε με την πρότασή μα. Δεν προτείνουμε να αλλάξουμε τους κανόνες, αλλά απλά και μόνο να βελτιώσουμε τα μαθητικά κείμενα και να απλουστεύσουμε τις τρέχουσες διοικητικές και νομοθετικές διαδικασίες. Η Κομισιόν καλωσορίζει τις περισσότερες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από την αξιότιμη εισηγήτρια ΔΕΛΑΕ που ακολουθούν τον ίδιο στόχο. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάποιες ανησυχίες για τις προτινόμενες αλλαγές όσον αφορά κάποια προϊόντα και τα μείγματα. Η αλλαγή των τωρινών κανόνων επιφέρει περισσότερη αυστηρότητα και περισσότερη απλότητα για τους εμπλεκόμενους. Επίσης, η απαγόρευση γλυκαντικών και συγκεκριμένα αλκοολούχα νομίζω θα επιφέρει σημαντικές δυσκολίες σε κάποιους εκπροσώπους του κλάδου. Η Κομισιόν επίσης καλωσορίζει την πλειοψηφία των τροπολογιών σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα. Όμως η προθεσμία των έξι μηνών χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση και πριν αναλάβουμε τέτοια δέσμευση θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν είναι σε θέση να τηρήσουν τις προθεσμίες. Καταρχάς, ο κανονισμός θα μπορούσε να καθορίσει το, την περίοδο ελέγχου στα πλαίσια της υπερκουρικότητας σε συνεργασία με τις χώρες μέλη και τους ελέγχους της Κομισιόν. Θα πρέπει να αποκλειστούν βεβαίω ε, πρόδειλα λάθιος όσον αφορά ε, τις προθεσμίες και επιπλέον οι τροπολογίες που αποβλέπουν στην εφαρμογή της αρχικής διαδικασίας δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα βάσιμες και θα πρέπει, θεωρεί η Κομισιόν, να υπάρχουν πιο ισόρροπα και αποτελεσματικά αποτελέσματα για όλο τον κλάδο των αλκοολούχων. Και στο πλαίσιο αυτό είμαστε στην διάθεσή σα να δώσουμε διευκρινήσεις και να απαντήσουμε ερωτήματα τα οποία μπορούν να ανακύψουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντελέ. Παρακαλώ πολύ σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σημείωσα κατά λεπτό στις ε, Παρατηρήσει των συναδέλφων. Φυσικά η γνωμοδότησή μου, το σχέδιο γνωμοδότησης αποτελεί μια βάση για τη συζήτηση και φυσικά ε, είμαι ευαίσθητη στα σχόλια των Ισπανών σε ό,τι αφορά την προσθήκη ζάχαρης. Θα φροντίσω λοιπόν ώστε η γνωμοδότησή μου να αντικατοπτρίζει τις εθνικές ευαισθησίες και να μην ε, είναι αφορμή να εκτεθούν διάφοροι κλάδοι σε επιμέρους χώρες σε δυσκολίες. Το αντίθετο θέλουμε να τους προστατεύσουμε, όχι να τους ε, πλήξουμε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τα θετικά του σχόλια. Διαπιστώνω πάντως ότι αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς θα πρέπει να είμαστε μέχρι τέλους και σε ό,τι αφορά την εξάμεινη προθεσμία που είναι η ευθυγράμμιση με την αντίστοιχη αναγνώριση που γίνεται για τα άλλα τρόφιμα, γιατί να μην έχουμε αντίστοιχη επίσπευση των εργασιών και για τα αλκοόλουχα ποτά, όπως ισχύει για τα υπόλοιπα τρόφιμα. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε, είμαι στη διάθεσή σας για συνέχιση των συζητήσεων και εγώ και οι συνεργάτες μου ε, προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι καθήλυνοι για το θέμα αυτό. Απλώς γνωμοδότηση συντάσσουμε, αρμόδια κατ' ουσίαν Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και εμείς είμαστε Επιτροπή Γεωργίας, όχι Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά και εσείς προσπαθήστε να μεταφέρετε αυτά τα σχόλια στην ομάδα σας, όπως κάνω και εγώ. Το γεγονός ότι ε, ε, συντάσσουμε απλώ γνωμοδότηση δεν σημαίνει ότι η δική μα γνώμη δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να, ότι δεν θα είναι αποφασιστική όσο και η έκθεση τη επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ώστε να ληφθούν υπόψη τα σχόλιά μα με πιέση προ του συναδέλφους. Ευχαριστώ. Προθεσμία για τι τροπολογίες ε, στι 14 Ιουλίου λίγη προθεσμία μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Παράμε στο επόμενο θέμα. Την παρουσίαση από τον κύριο Χόσλινγκ των αποτελεσμάτων του τριμερούς διαλόγου για τα βιολογικά προϊόντα. Ευχαριστούμε θερμά και την κυρία Μπενίτες Σάλας. εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας έχουμε ε, ενημερώσει σχετικά και με γραπτά σημειώματα, οπότε ε, ε, περιμένουμε πρώτα το πράσινο φως από το Συμβούλιο για να εγκρίνουμε το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου, οπότε ε, πρέπει να περιμένουμε το φθινόπωρο, δηλαδή την επάνωδό μας μετά τις θερινές διακοπές. Ο κύριος Χόισλιν θα μας ενημερώσει. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί και οδησυγητές. Όντως, μετά από 20 ολόκληρους μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων και κατά τη διάρκεια του 18ου τριμερούς διαλόγου, καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για ένα κείμενο για το οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι, όχι επειδή είναι τέλειο, υπάρχουν ακόμα κάποια σημαντικά σημεία τα οποία θα πρέπει να αποσαφινιστούν μέσω κατεξότηση πράξεων στο εγγύς μέλλον, αλλά επειδή το κείμενο τελικά αυτό αντικατοπτρίζει πολλά διαφορετικά συμφέροντα τα οποία πρέπει να ενταχθούν τελικά στο ίδιο πλαίσιο. Υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία για διάφορους λόγους δεν έχουν καλυφθεί εντελώς, αλλά πάντα αυτό συμβαίνει στα πλαίσια ενός συμβιβασμού. Έπρεπε να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση, προκειμένου να μην στραφούμε κατά της ε, γεωργικής ανάπτυξης τελικά. Να σε ευχαριστήσω λοιπόν όλους για την υποστήριξή σας, την υπομονή σας, την επικοδομητική σας συνεργασία. Σίγουρα ήταν με πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, 20 μήνες, τέσσερις ολόκληρες προεδρίες του Συμβουλίου προσπάθησαν να συγκεράσουν τις διαφορετικές αυτές απόψεις που ακουγόντουσαν στα πλαίσια του Συμβουλίου και τελικά μόνο η Μαλτέζικη Προεδρία τα κατάφερε στο τέλος. Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέδειξε επικοδομητική στάση. Μας υποστήριξε, ήταν σε θέση πάντα να κάνει συμβασμούς. Θα, θα λοιπόν ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στάση που κράτησε. Και βέβαια να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις συγητές εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δική τους την υποστήριξη χωρίς την υποστήριξή σας τίποτα δεν θα είχε πραγματοποιηθεί. Τα καταφέραμε λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σημειώσουμε πρόοδο σε πάρα πολλά από τα σημεία τα οποία θέλαμε να προωθήσουμε. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους συναδέλφους. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος εργασίας έγινε από τη γραμματεία μας και από το προσωπικό της γραμματείας μας. Και Όλε οι πολιτικέ ομάδε θεωρώ συνέβαλαν πάρα πολύ σημαντικά του τελευταίου αυτού 20 μήνε. Για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ όλου πάρα πολύ. Το συμβούλιο που θα λάβει η χώρα τον Ιούλιο θα εγκρίνει το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων, τη σημαντική αυτή λύση και θα πρέπει να γίνει ακόμα μια τεχνική εργασία στα πλαίσια τη Εστονική Προεδρία. Εμεί τώρα στη δική μα την Επιτροπή θα σας παρουσιάσουμε το κείμενο προς έγκριση κατά πάσα πιθανότητα τον Οκτώβριο και μάλλον θα πάμε σε μια ολομέλεια προς τα τέλη του 17 στις αρχές του 18. Και αν όλα πάνε καλά, το 2020 θα τεθεί, θα ο κανονισμός αυτός. Πολλά πράγματα νομίζω ότι ήδη έχουμε πει ως προς το περιεχόμενο του κανονισμού, ας πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι με το τελικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λίντσε για μια σύντομη παρακαλώ ε, παρουσίαση. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ επικοδομητική συνεργασία που είχαμε. Ο κύριος Σάουσλινγκ είπε ότι ο ε, συνήθω στα πλαίσια της πολιτικής διαδικασίας πρέπει να καταλήγουμε σε μια συμβαστική λύση που βέβαια δεν είναι πάντα ιδανική για όλους τους εμπλεκομένους, αλλά μην ξεχνάμε το σημείο θετηρίας. Οι περισσότεροι εξημών θέλαμε να μην έχουμε τις ε, οριακές αυτές τιμές ε, το που πρότεινε το Συμβούλιο όσον αφορά τα ζανιοκτώνα. Θέλαμε πιο αυστηρά ανώτατα όρια, θέλαμε πιο αυστηρούς ελέγχους, καλύτερο σύστημα επιτήρησης. Όλα αυτά τα πετύχαμε, καταφέραμε να τα διασφαλίσουμε στο τελικό κείμενο. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο χαίρομαι πάρα πολύ που πολλοί βλεκόμενοι από τον κλάδο, από την Κόπα Κοζέκα για παράδειγμα ή από άλλες οργανώσεις έχουν ήδη χαιρετήσει πολύ θετικά το τελικό αυτό κείμενο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η συμβαστική αυτή λύση όντω διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή οικονομική ανάπτυξη αυτού του κλάδου. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Αντριέ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ, όπως και ο Νόρμπερτ, να εκφράσω την ευαρέσκειά μου για το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης και να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας τον κύριο Χόισλινγκ που κατάφερε και πέρασε το φιλοπορίας που είχαμε εκπονήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρά τη μακροχρόνια και επίπονη προσπάθεια των τριμερών διαλόγων. Πάντως, ε, είχαμε αγαστή συνεργασία με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και με τις δικές μας υπηρεσίες και καταλήξαμε σε μια συμβαστική λύση που θα μας επιτρέπει να ανταπεξέλθουμε στις τεράστιες προκλήσεις και στα διακυβεύματα. Ήσασταν και εσείς στους τελευταίους τριμερείς διαλόγους και είδατε πόσο περίπλοκο είναι το θέμα ε, και άπτεται πολλών ε, γεωργικών κλάδων. Είναι οριζόντιο. Σε θέματα ελέγχου και για τις τρίτες χώρες καταλήξαμε σε μια ενδιαφέρουσα συμβαστική λύση που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε. Το ίδιο και για τις όρους προσπορά και για τα κατόφλια. Νομίζω ότι τα θεσμικά όργανα ε, αντελήφθηκαν τη, τις ευθύνες τους ε, και θεωρώ ότι ε, καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε στο ύψος των περιστάσεων και των διακυβευμάτων με την συμβαστική αυτή πρόταση. Ο κύριος Ντόρφμαν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δυστυχώς ε, δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτή την αγαλίαση και την γενική εφορία. Ε, δυστυχώς σε κέρια ζητήματα δεν καταφέραμε να καταλήξουμε συμφωνία και όπως είπα και στο παρελθόν ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην ουσία και αυτό ισχύει για τα κατάλοιπα για παράδειγμα των φυτοφαρμάκων. Και μάλιστα πολλές ενός και οργανώσεις μας το επισήμαναν όταν το κοινό μάθει ότι ακόμη και βιολογικά τρόφιμα μπορεί να φέρουν κατάλοιπα φυτοφαρμάκων αντίστοιχα με τα προϊόντα της συμβατικής γεωργίας θα αρχίσουν να διαρωτώνται πού πήγε στραβά το θέμα. Εγώ δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένο με τη συμβαστική πρόταση. Ο κύριο Ταραμπέλα. Ε, χαίρομαι για το σχόλιο του κύριου Ντόρφμαν, γιατί νομίζω ότι ήταν φιλόδοξο αρχικά ο στόχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ό,τι αφορά τη βιολογική παραγωγή και πραγματικά ο κλάδο θα ένα αυστηρότερο κανονισμό για να τον προστατεύσουμε, γιατί είναι ένας ε, ε, τομέα που ακμάζει με αυξανόμενη ζήτηση και γι' αυτό θα έπρεπε να τον προστατεύσουμε καλύτερα. Για τους πόρους προσφορά ήταν τεράστια η πρόοδο ό,τι αφορά του προσωρινού πειραματισμού, τη βιολογική παραγωγή και το γεγονό ότι κάποιε πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον ενώ ε, απαγορεύονται σήμερα. Εξαίρεση και για τη βάση δεδομένων. Θετικό. Έλεγχο των εισαγωγών. Είναι σαφέ ότι το σημείο αυτό ήταν σημαντικό και πραγματικά η πρόοδο αρκετά εντυπωσιακή. Αντίθετα, σε ό,τι αφορά τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων, εκεί ήταν κέριο το ζήτημα. Έπρεπε να επιδιώξουμε μια εναρμόνιση και, καταλήγουμε σε, και να καταλήξουμε σε ένα κανονισμό που να ισχύει παντού στην Ευρώπη. Δυστυχώ δεν ε, υλοποιήσαμε τι φιλοδοξίε ε, ε, όσο αφορά του κανόνε βιολογική παραγωγή για τους ελέγχους. Μερικές φορές είναι αιτήσιοι, άλλες φορές κάθε δύο χρόνια ένας ε, τομέας που ακμάζει προσφέρεται και για πάτες, όχι υπερβολικούς ελέγχους λοιπόν, αλλά έπρεπε να εξασφαλίσουμε επαρκείς ελέγχους για να αναχαιτήσουμε τις απάτες και την παραγωγή ε, εκτό εδάφου ε, χωρίς χώμα. Είναι αρκετά ελαστικό αυτό το θέμα, αρκετά ευελιξία. Θα πρέπει να όμως να ισχύει για τη βιολογική παραγωγή η βασική αρχή του συνδέσμου με το χώμα, με τη γη. Δεν συμμερίζομαι λοιπόν τον υπέρμετρο θυσιασμό που έδειξε αυτό ο σκόπος ε, για να καταλήξουμε σε ένα προβληματικό κανονισμό. Ο κύριος Χόσλινγκ ε, ήταν πράσινος. Ήλπιζα να είχαμε έναν ε, κανονισμό που θα προστατεύει πραγματικά τη βιολογική παραγωγή. Προστατεύει μεν τη βιολογική παραγωγή, αλλά στους μεγάλους επιχειρηματίες ει βάρος των μικρών καλλιεργητών και νομίζω ότι το σήμα που θα εγκρίνουμε τον κανονισμό θα αποβεί εις βάρος των μικρών βιολογικών καλλιεργητών. Εγώ δυστυχώς δεν θα μπορέσω να υπερψηφίσω τον κανονισμό όποια και αν είναι η επίσημη θέση της ομάδας μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Νόιχλ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ ή ότι συμφωνώ λιγότερο ή περισσότερο. Δεν ξέρω. Πάντως δεν το έχω δει το κείμενο ακόμα. Πάντως να αναφερθώ στους 20 μήνες διαπραγματεύσεων για το κατά πόσο κάποιο θα εδώ ή όχι ε, δεν είναι και τόσο σημαντικό, αλλά ούτω ή άλλω 20 μήνε ήταν πολύ μεγάλη περίοδο, πολύ μεγάλη προθεσμία για τον κλάδο. Πολλά πράγματα καθυστέρησαν, ιδιαίτερα στον τομέα των βιολογικών και είδαμε τι ζημιά έχει αυτό. Είδαμε οργανώσει ε, βιολογικών παραγωγών στη Γερμανία μα έλεγαν μην το υπογράψετε, αλλά μα έλεγαν υπογράψτε το. Οπότε ε, τα πράγματα ήταν ή έγιναν πάρα πολύ δύσκολα όσον αφορά τα βιολογικά. Όταν λέει ο κόσμος ότι αυτό αποτελεί ένα σημείο καμπής, μπορεί να είναι είτε αρνητικό είτε θετικό. Οπότε θα πρέπει να το εξετάσω προσεκτικά. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα συστήσω η ίδια στην ομάδα μου σε σχέση με την ψηφορία. Πάντως έχω συγκεκριμένες και πολύ σοβαρές στάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, μόλις παρατήρησα βλέποντας τη σύνοψη της έκθεσης ότι το λόμπι των βιολογικών θα ήθελε να σταματήσει να αποτελεί ένα περιορισμένο κλάδο. Αλλά νομίζω αυτό ακριβώς τους βοηθάει. Γιατί αν δεν είναι κάποιος εξειδικευμένος ε, κλάδος γίνονται κάτι το καθημερινό. Και φαίνεται ότι θέλουν να αφαιρέσουν όλα τα όπλα των φαρμάκων. Οπότε, αν κάποιος θέλει να τα αφαιρέσει όλο και περισσότερο, τότε γιατί κάποιος να αγοράσει βιολογικά. Επίσης, οι απάτες. Είναι πολύ εύκολο να βάλουμε σήμανση βιολογική, αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις κιόλας τι αγοράζεις μπορεί να φωνάζουν η παραγωγή βιολογικών ε, προϊόντων, ξέρω εγώ, για την ποιοσιμότητα. Είναι όμω να, να παίρνουμε, να εισάγουμε βιολογικά από την Ρουμανία. Οπότε θεωρώ ότι η παραγωγή βιολογική θα πρέπει να είναι τοπική και η παραγωγή θα πρέπει να έχουν ακριβώ και λόγο στι αποφάσει που του αφορούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της, την εκπρόσωπο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Μπενίτα Σάλλας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Κομισιόν, όπως είπατε κι εσείς, αρχικά είχε ένα πολύ πιο φιλόδοξο στόχο. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις ουσίες που επιτρέπονται ή όχι. Όμως, Πρόεδρε, η καλύτερη συμφωνία δεν είναι αυτή που περιλαμβάνει την τάδη ή ρήτρα, αλλά αυτή που μπορεί να υπογραφή και που κάνει μια κατανομή ισομερή της αποδοχής και της απόρριψης. Το θέμα αυτό είναι αρκετά περίπλοκο και ε, τελικά καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό και να επιμείνω για το ότι το γεγονό και μόνο ότι καταλήξαμε σε συμβασμό έστω και αν αυτός δεν είναι τέλειος ήδη καταδεικνύει τη δυνατότητα διαπραγμάτευση εκ μέρου των θεσμικών οργάνων. Θα ήταν χειρότερο για το κλάδο των βιολογικών και όχι μόνο για τα βιολογικά, αλλά γενικότερα για του θεσμού. Πέρα από το καθαρά γεωργικό στοιχείο, θα ήταν πολύ αρνητικό να αποδείξουμε στην κοινωνία ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για τα απλά, για ένα απλό συμβασμό. Τώρα, τούτο λεχθέντος θεωρεί η Κομισιόν ότι βρίσκεται στα όρια της δικαιοδοσία της και των ομοιοτήτων της η εντολή αυτή, λέει η Κομισιόν, πιστεύει η Κομισιόν και θεωρούμε ότι το αποδεχόμαστε επειδή ακριβώς παρέχει κάποια πλεονεκτήματα όπως το να περάσουμε στις διεθνείς συμφωνίες από την αντιστοιχεία στην συμμόρφωση, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους ε, παραγωγούς που τους βάζει σε ισότιμους όρους ανταγωνισμού με παραγωγούς τρίτων χωρών. Οι έλεγχοι, οι κατά την άποψή μας δεν υποχωρούν, δεν εξασθενούν το αντίθετο, γιατί μπορούν να ενισχυθούν σε μέρη και, και περιοχές όπου πραγματικά υπάρχει κίνδυνος ώστε να έχουμε καλύτερο έλεγχο. Θεωρούμε λοιπόν, α, μάλιστα, επίση να τονίσω ότι βάσει του κανονισμού που ισχύει αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν δυνατόν να κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε, θα μπορούσαμε να εκθετήσουμε νέου κανόνε που θα συνοδεύουν αυτόν τον τόσο δυναμικό τομέα στην ανάπτυξή του, όπω είπατε και εσεί. Γιατί, γιατί ο τωρινό κανονισμό δεν έχει αβωνοποιηθεί. Οπότε δεν θα είχαμε κάποια βάση για να δράσουμε. Οπότε καλωσορίζουμε το συμβασμό αυτό και ελπίζουμε να υιοθετηθεί μέσω της διαδικασίας λεψοφάσεων της συνήθους των θεσμικών οργάνων και να μπορέσουμε να το υπογράψουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Χόισλιν και πάλι ο εισηγητής ίσως πρέπει να δευτερολογήσει. Κυρίες και κύριοι, ε, όταν μιλούμε για συμβαστική λύση εξορισμού δεν μπορεί να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Και ακριβώς ε, εκεί έγκυται ο καλός συμβασμός όταν ε, κανείς δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένο, όλοι έχουν κάνει υποχωρήσεις. Ξέρουμε ποια είναι η θέση του Συμβουλίου, ποια είναι η θέση των οικολόγων και των παραγωγών βιολογικών προϊόντων. Είναι εξαιρετικά περίπλοκο το θέμα και νομίζω ότι το γεγονό ότι καταλήξαμε συμβασμό δεν είναι κακό. Κύριο Χόισλινγκ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Να σας δώσω και τα συνδευτικά έγγραφα α, να δείτε πόσο περίπλοκο ήταν και σα έχω και καλέ διακοπές κιόλα. Να δείτε πόσο δύσκολο όχι ήταν να, πόσο δύσκολο ήταν όχι να καταλάβουμε τα περίπλοκα, τα δύσκολα ζητήματα, αλλά τα βασικά, τα απλά. Και στο Συμβούλιο είχαμε μία απόψη απόψεων 50-50 Οπότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Οπότε είπαμε να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα συμβασμό, να το βάλουμε κάτω και να συζητήσουμε και να δούμε ακριβώς και την έκθεση της Κομισιόν σε σχέση με το από πού προέρχεται η μόλυνση. Πάντως θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε στο πλαίσιο των νέων κανονισμών που έρχονται και η νομοθετική διαδικασία είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να ενσωματώνουμε νέα δεδομένα και νέες πληροφορίες όσο αυτά ανακύπτουν. Με τις διαπραγματεύσεις αυτές, σε δύο περιπτώσεις κοντέψαμε να αποτύχουμε γιατί το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να καταλήξει συμφωνία και υπό ο Μαλτές και η Προεδρία την τελευταία στιγμή βρήκαμε κάποια συμφωνία και συμβασμό. Οπότε θα ήθελα να το πω αυτό προς τους αδέλφους που είναι επικριτικοί ότι τι θα ήταν ε, η άλλη εναλλακτική το να μην έχουμε καθόλου κανονισμό. Τουλάχιστον εδώ έχουμε ένα κανονισμό που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε. Το χειρότερο για το σύνολο της Ένωσης θα ήταν να μην έχουμε τίποτα. Τουλάχιστον εδώ έχουμε ένα συμβασμό. Οπότε Ξαναλέω, είχαμε πάρα πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις και μπορέσαμε να έχουμε τουλάχιστον αυτό το συμβασμό που προσφέρει κάποια προστιθέμενη αξία σε σχέση με τον κανονισμό που ούτως ή άλλως θα έπρεπε να αλλάξει. Οπότε ξαναλέω τι είναι καλύτερο αλλαγή του παλαιότερου ή του νέου κανονισμού, δεν ξέρω. Αλλά τέλο πάντων τουλάχιστον έχουμε κάτι τώρα στα χέρια μα, κάτι το αυτό. Και μάλιστα ξέρω ότι στη Γερμανία πάρα πολλοί δεν ήθελαν νέο κανονισμό. Και ε, έπρεπε να τους πείσουμε ότι θα ήμασταν καλύτερα με ένα νέο κανονισμό αντί με τον παλαιότερο. Τέλος πάντων, ε, να το ξανασυζητήσουμε αν θέλετε, αλλά εγώ ξαναλέω αυτά που είπα προηγουμένω και νομίζω ότι αυτή είναι και η άποψη των συναδέλφων που συνδιαπραγματεύτηκαν μαζί μου, ότι το Κοινοβούλιο πέτυχε κάτι το οποίο νομίζω μπορεί και πραγματικά μας κάνει περιπέτεια. ευχαριστώ πολύ. Εγώ προσωπικά, έχοντας παρακολουθήσει και το τέλος των διαπραγματεύσεων, θεωρώ ότι περισσότερες υποχωρήσεις για τη συμβαστική λύση έκαναν το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λιγότερες υποχωρήσεις έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. λάβατε το παρακαλώ και αυτό υπόψη. Πάντως η διάσταση απόψεων υπήρχε σε όλα τα θεσμικά όργανα ούτω ή άλλω. Ευχαριστώ θερμά. Μπράβο σα κύριε Χόισλινγκ. Πραγματικά αργόδης προσπάθεια χρονοβόρα διαδικασία, μακροχρόνιε εργασίε και α έχουμε τελικά, α ελπίσουμε ότι θα έρθει σε αίσιο πέρας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους ε, για την συμβολή τους ε, στην ε, αίσια διεκπαιρέωση του τριμερούς διαλόγου. Μας έμεινε ένα θέμα, έχουμε 8 λεπτά ακόμη διερμηνία. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Ντές που θα μας ενημερώσει για την πορεία των τριμερών διαλόγων για το Omnibus. Αν δεν προλάβουμε σήμερα μπορούμε να συνεχίσουμε και αύριο πάντως. Κύριε Ντές παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι, για το Omnibus. Να σας πω ότι μπορέσαμε να καταθέσουμε έγκυρα τη θέση μας. Είχαμε τον πρώτο τριμερή και την πρώτη συνάντηση των σκιωδών και θα ξανασυστήσουμε σε αυτά του Σεπτέμβρη. Ο πρώτος τρεμερής στις 5 του Ιούλη πήγε καλά. Κοιτάξαμε ακριβώ εκεί τα οριζόντια ζητήματα και την ΚΟΑ για τον οριζόντιο κανονισμό. Να πω τα εξή, Εδώ θα πρέπει να δούμε ακριβώ τι γίνεται με τα προβλήματα που αφορούν την εθνική και την, και, την κοινωνική νομοθεσία σε τεχνικό επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Είχαμε επίσης το θέμα του 4% το οποίο δεν έγινε δεκτό στα πλαίσια του προπολογισμού. Είχαμε και το έτοιμο του Κοινοβουλίου για το αποθεματικό για περίπτωση εκτακτής ανάγκης. θεώρησε η νομική υπηρεσία ότι αυτό αποτελούσε έτσι, κάποιο, ότι παρουσίαζε κάποιο πρόβλημα επειδή δεν είχε ακολουθεί η σωστή διαδικασία. Και από το 4 που είμαι στο Κοινοβούλιο βλέπω εγώ να ζητάμε συνεχώς το αποθεματικό να αυξάνεται αλλά δυστυχώς αυτό δεν γίνεται δεκτό. η Κομισιόν και το Συμβούλιο συμφώνησαν με το Κοινοβούλιο. Θα υπάρξει ακόμα μια τεχνική συνάντηση. Θα μιλήσουμε για το πακέτο 4, τα συστήματα ελέγχου. Έχουμε και την τροπολογία 360, όπου ακριβώς έχουμε την ίδια θέση για το Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο και η Συμφώνηση Κομισιόν. 5. Για το 5 η Κομισιόν θα προετοιμάσει μια δήλωση που θα συζητηθεί στην Τεχνική Επιτροπή για να δούμε ακριβώς κατά πώς το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να συμφωνήσει και αυτό. Στο Κοινοβούλιο εμείς πάντως πήγαμε παραπέρα, πιο πέρα από το Συμβούλιο, το οποίο ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τις συζητήσεις του. Οπότε θα χρειαστεί και η επόμενη εβδομάδα, αλλά μέχρι τώρα το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να μας μεταβιβάσει τη θέση του επειδή ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί και συνεχίζουν εσωτερικά τις συζητήσεις. Για τα φρούτα, τα όσπρια και τον ίνο αντίθετα έχουμε καταλήξει σε συμφωνία. Ήταν το πρώτο αποτέλεσμα του τρομερούς ε, διαλόγου. Ευχαριστώ και τον Σάλφο Δεκάστρο που συνεργάστηκε μαζί μα και που μας παρουσίασε τη θέση του Κοινοβούλου. Ευχαριστώ. Ο κ. Δεκάστρο. Ε, τα είπατε όλα, τα είπατε όλα συναλφεντές. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να πω ότι ήταν κάπως δύσκολο αυτό το Συμβούλιο γιατί σε, πολλές, σε πολλά ζητήματα δεν είχε θέση. Οπότε ε, εύχομαι την επόμενη εβδομάδα με το Συμβούλιο Γεωργίας και με το ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πάντως καταγράφω σημαντικά πράγματα πρόοδου της Κομισιόν που μας χαροποιούν αλλά στις 7 του Σεπτέμβρη και στις 24 θα έχουμε τους σημαντικούς τριμερείς. Ελπίζουμε εκεί να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σύντομα και να καταλήξουμε στον τελευταίο τριμερή στις 14 του Οκτώβρη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Βλέπετε, στείλαμε στην πρώτη γραμμή του πυρός ε, πολύ πεπειραμένους μαχητές εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος κάνω παρακαλώ. με κάθε σεβασμό. Γιατί το τελευταίο σημείο το παραμαζεύουμε συνεχώς. Δεν μπορούμε να ξεκινάμε εγκαίρως ε, τη συνεδρίαση. Θα είχαμε ένα 20 λεπτό αν είχαμε ε, ξεκινήσει έγκαιρα. Αλλά έφυγε και δεν μ' άκουσε. <laughs> Κύριε Πρόεδρε, Ενδεχομένως ε, να μην είναι αναγκαίο να κάνουμε εδώ μια εκτενέστατη συζήτηση. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε τριμερή διάλογο άλλωστε για το ζήτημα αυτό. Ακούσαμε διάφορες εξηγήσει για τις τροπολογίες. Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες είτε πειράζουν τον προπολογισμό αυτό καθεαυτό είτε όχι. Το πιο σημαντικό για μας είναι ότι το Συμβούλιο πρέπει γρήγορα να καταλήξει σε μια θέση προκειμένου να ασχοληθούμε με το περιεχόμενο της θέσης του Συμβουλίου. Να σας ευχαριστήσω πάνω για τη συζήτηση που έχει γίνει μέχρι τώρα. Νίκολσον, πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με τους το πιο σημαντικό είναι να δούμε ότι δεν υπάρχει θέση του Συμβουλίου. Αυτό μα αγανακτεί βέβαια αυτή τη στιγμή. Εμεί είμαστε έτοιμοι να κάνουμε βήματα πρόοδου. Α δούμε τι θα κάνει και το Συμβούλιο από τη δική του την πλευρά. Δεν ζήτησε άλλο κανεί το λόγο. Οπότε θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Μίχαελ Νιέγιαρ, από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργία. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σα. Θα ήθελα απλώ να ευχαριστήσω του συμμετέχοντε στον τριμερή διάλογο. Νομίζω ότι σημειώσαμε αρκετή πρόοδο για του δύο κανονισμού και στον επόμενο τριμερή διάλογο θα δούμε τα εκκρεμή ζητήματα ώστε να διαμορφώσουμε μια πλήρη εικόνα και ευελπιστώ ότι θα βρούμε κοινά σημεία για συμβαστική λύση για τον κανονισμό Omnibus. Εμείς Είμαστε υπέρ μια επικοδομητική συνεργασία. Αυτή ήταν η στάση μα και μέχρι στιγμή. Αλλά μα πιέζει το χρονοδιάγραμμα. Γιατί μέχρι τι 12 Οκτωβρίου, που είναι η τελευταία ημερομηνία του ημέρου διαλόγου, θα πρέπει μέχρι τότε να διεκπαιρεώσουμε το θέμα αυτό. Ναι, να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο κύριο Ντε. Ότι ε, και ο κύριος Δαντά συνέβαλε ε, στην πρόοδο των εργασιών. Ο κύριος και πάλι. Σας ευχαριστώ. Ήθελα απλώς να πω κάτι για τις επικρίσεις που ακούσαμε. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε αρκετό χρόνο στην Επιτροπή Γεωργίας για να συζητήσουμε εκτενώς το θέμα αυτό. Και ε, εξεπλάγει από τη δυσκολία του Συμβουλίου να καταλήξει εκείνη η θέση ε, Εμεί είμαστε μια ολιγομελή ομάδα και καταφέραμε πολύ γρήγορα να καταλήξουμε σε θέση, αλλά τα εθνικά υπουργεία έχουν πολλού υπαλλήλου, γι' αυτό δεν είναι εύκολο το Συμβούλιο να καταλήξει. Ναι, καταλήξαμε σε πρόταση, αλλά οι δικέ μα προτάσει δεν είναι καθόλου εύκολε για το Συμβούλιο. Οπότε έχει νόημα το, το Συμβούλιο να σκεφτεί εκτενώς τις προτάσεις μας που παραλαμβάνω θα είναι δύσκολες να τις αποδεχτεί το Συμβούλιο. Το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή στην απογευματινή συνεδρίαση κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει ο για τα επιπλέον λεπτά που μας παρήχαν. Καλό σας βράδυ. Ραντεβού αύριο στις 9 το πρωί. Γεια σας.